Okay, good morning everybody. Καλημέρα σας. Θα ξεκινήσουμε την ψηφοφορία τώρα. Δυστυχώς με μία μικρή καθυστέρηση. During... Ε, κανονικά μιλάω σου αλλά για την ψηφοφορία νομίζω ότι θα είναι ευκολότερο εάν ε, μιλούμε <clears throat> αγγλικά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα την συνεδρίαση ε, με το σημείο υπαριθμών 11 της Μερισίας Διατάξεως σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2012. Maybe Μήπως θέλετε το λόγο για προφορική τροπολογία, ναι. Σχετικά για την τροπολογία 7, δεν ξέρω εάν θέλετε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία και να μιλήσω για το θέμα αυτό όταν έρθει... Ε, α, τώρα? Εντάξει. Τροπολογία 7 λοιπόν επί της παραγράφου 23. Προφορική τροπολογία ε, που θέλει να αντικαταστήσει τρεις λέξεις social automatic stabilizers αυτό να αλλάξει και να γίνει they. Αυτές οι τρεις λέξεις λοιπόν να αντικατασταθούν από την ε, αντωνυμία αυτή. Οι σταθεροποιητές. Αυτό ήθελα μόνο. Αντικατάσταση των τριών λέξεων με το they στα αγγλικά. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι από τις τροπολογίες 1 έως 6 δεν υπάρχει αντίθετη γνώμη, επομένως μπορούμε unblock όχι. Εντάξει, μία προς μία λοιπόν θα τις ψηφίσουμε. Okay, so take one to three block. Unblock 1, 2, 3. Ούτε δεν πειράζει. Μία προς μία λοιπόν, κανένα πρόβλημα. Okay, we start with Amendment 1. Now you see me. And uh, Those are... Υπέρ της πρώτης τροπολογίας κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Α, συγγνώμη, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. Ναι, τροπολογία 5, 5, τροπολογία 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 και μετά έχουμε μια προφορική, επ' έχουμε προφορική τροπολογία. Ε, υπάρχει αντίρρηση σχετικά με την αποδοχή αυτής της προφορικής τροπολογίας. Όχι, άρα ψηφίζουμε. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 8, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές ναι, νομίζω ότι εδώ πρέπει να κάνουμε επαλήθευση. Ωραία, ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Ναι, εγκρίνεται τελικά. 12 and 12. Σημείο 12 της μερισσίας διατάξεως, ενεργειακή απόδοση. And we first start with amendment number... Τροπολογία 14. Υπέρ. Παρακαλώ, να σηκώνετε τα χέρια σας. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. <clears throat> Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 έχει αποσυρθεί, άρα τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρα και η τροπολογία 7 καταπίπτει. Όχι. Τροπολογία 7. Την ψηφίζουμε κανονικά. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 11 και εδώ έχουμε ψηφοφορία κατά τμήματα που έχει ζητήσει το ΕΛΚ. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι θα πρέπει να το ελέγξουμε. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Για την τροπολογία 13 ψηφίζουμε. The vote is closed. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε τώρα επί του τροποποιημένου κειμένου με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. And vote is now closed. Και εγκρίνεται. Και συγχαρητήρια βεβαίως στην εισηγήτρια. then moving on to item 13, the Daphne program, and I will first... περνούμε τώρα στο ε, σημείο 13, το πρόγραμμα Δάφνη και το λόγο έχει η κυρία Πάστος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδης ηγητές με τους οποίους συνεργάστηκα πάρα πολύ καλά Ε, θα μπορούσα να αναφέρω όλα τα ονόματα, αλλά θα αναφέρω μόνο την κυρία Κιγιώμη, η οποία μπλοκαρίστηκε από τις απεργίες ε, στη Γαλλία. 73 είναι οι τροπολογίες που κατατέθηκαν, συνενετικές οι περισσότερες, ορισμένες ε, ε, είναι καινούριες ιδέες. Η δική μου μέρημνα ήταν να ενισχύσουμε τη χρηματοδότηση του προγράμματος Δάφνη το οποίο εντάσσεται σε ένα πιο ευρύ πρόγραμμα ε, ε για την περίοδο 2014-2020 και πέραν αυτού, ε, πέραν της ένταξης σε ένα πιο ευρύ πρόγραμμα, προσπαθούμε να μην χάσει την παρουσία του, την ορατότητά του, γιατί είναι πολύ σημαντικό στον αγώνα κατά τη ε, βία εναντίον των γυναικών, των νέων και των παιδιών. Αυτή ήταν η βασική μέρημνά μου και όλων μας. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία και ιδιαίτερος ευχαριστώ τη γραμματεία της ε, Επιτροπής ε, για την πολύτιμη βοήθειά της. Ευχαριστώ. we don't Λοιπόν, περνούμε στην ψηφοφορία. Αρχίζουμε με την τροπολογία υπαριθμών 23. Παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σημαίνει ότι 24 καταπίπτει. Συμβαστική. πίνει υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι 31, 32, 29, 27, 26, 30, 28 και 25 καταπίπτουν. Ε, συμβιβαστική 4. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τούτο σημαίνει 33 πίπτη. Τροπολογία 34. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τούτο σημαίνει ότι η τροπολογία 35, 40 και 38 καταπίπτουν. Περνούμε στην 36. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Περνούμε στην 37. Ποιοι είναι υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 41, ε, 42, συγγνώμη, ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 43. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Να ελέγξουμε τη 42 παρακαλώ. Α, συγγνώμη δεν το άκουσα. Ωραία. Ελέγχουμε την 42 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 42 παρακαλώ. Has everybody voted? Ψηφίσατε άπαντες. Now, the vote is closed. Πέρας. Απορρίπτεται, έτσι δεν είναι, ναι, απορρίπτεται. Μπορούμε να επανελέγξουμε παρακαλώ. Τώρα ψηφίζουμε τη 44. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45, 48, 47, 46 καταπίπτουν. Περνούμε στην 49. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50 και 54 από κοινού. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία υπαριθμών 51 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και 53 καταπίπτει και περνούμε στην 55. Α, έχει αποσυρθεί. Ακριβώς. Ε, πηγαίνουμε στην συμβαστική υπαριθμών 5. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται 62, 61, 57, 58, 60, 59 καταπίπτουν και περνούμε στην 63 ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική υπαριθμών 6 α θέλετε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά ωραία Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία υπαριθμών 63, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική υπαριθμών 6. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τούτο σημαίνει ότι οι 64 και οι 66 καταπίπτουν και ψηφίζουμε την 65. Υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Έχουμε τώρα την 67 και μια προφορική τροπολογία. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση, όχι. Μπορούμε να ψηφίσουμε λοιπόν την προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 68 καταπίπτει και ψηφίζουμε την 69. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 70 καταπίπτει. 71 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 72 καταπίπτει. 73 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία αριθμών 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 4 παρακαλώ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμών 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τούτο σημαίνει ότι οι τροπολογίες 8 και 7 καταπίπτουν. Τροπολογία υπαριθμών 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 11 καταπίπτει, 12 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 13. Ε, ε, τροπολογία 14 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία υπαριθμών 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 21 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 22 καταπίπτει και ψηφίζουμε την 1. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Και τώρα θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά το σύνολο του ψηφίσματος και άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Thank you very much. Κυρία Πάστο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Okay, we... Ωραία, λοιπόν. Και τώρα συνεχίζουμε τη συνεδρίαση και θα περάσω στα Σουηδικά. Ε, Ωραία, παρακαλώ. Συνεχίζουμε και θα περάσω στα σουηδικά. Eh, λοιπόν, συνεχίζουμε. Παρακαλώ να λάβετε τις θέσεις σας. Ε, παρακαλώ να βάλετε τα ακουστικά σας γιατί θα καταλάβετε τίποτα από όσα έχω να σας πω. Θα μιλήσω σου ειδικά. Μιλάω σου ειδικά τώρα. Και περνούμε στο σημείο 14 της ημερησίας διατάξεως. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω έχει καθυστερήσει η κυρία Πιέτη Κάινεν Ε, άρα θα πάμε στο σημείο 5. Παρακαλώ, αν θέλετε να συνομιλήσετε μεταξύ σας, παρακαλώ να το κάνετε εκτός αιθούσης. Ευχαριστώ πολύ. Λέει ο πρόεδρος. We don't λοιπόν, δεν μπορούμε να συζητήσουμε το σημείο 14, διότι δεν είναι παρούσα η συγγήτρια. Πηγαίνουμε στο σημείο 5, γυναίκες και κλιματική αλλαγή και θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια κυρία Κιλ Νίλσαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι τελικά φτάσαμε σε μια συμφωνία πιο φιλόδοξη που ε, μας ενθουσιάζει παρόλο που δεν είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα έχουμε δύο σημαντικά μηνύματα πρώτον για την Ευρωπαϊκή Ένωση χάρη στο έργο της ε, Επιτρόπου Έντγκαρτ άρχισε να, διαδρα... να συνεχίζει το ρόλο της, της ηγέτιδος στην κλιματική ε, πολιτική για την καταπολέμηση των όσων συμβαίνουν σε σχέση με την αλλαγή ε, του κλίματος. Πράγματι διαφοροποιείται η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείε και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή με τις δράσεις μας λαμβάνοντας υπόψη και τι προκλήσει τις προκλήσεις όσο και την, ε, το δίκαιο σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεύτερο μήνυμα. Οι γυναίκες βρίσκονταν σε θέση κλειδί, αν θέλετε, σε σχέση με αυτή την ε, συμφωνία. Τόσο σε σχέση με την Επίτροπο όσο και την Πρόεδρο, την Μάισε Καταμπάνα αλλά και την Κριστιάνα Φιγκέρες. Αλλά επίσης και σε επίπεδο μη κυβερνητικών οργανώσεων και παράλληλων δραστηριοτήτων. Οι γυναίκες συνεισέφεραν με τις γνώσεις και την εξειδίκευσή τους όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Δηλαδή οι γυναίκες εμφανίστηκαν ως ε, κεντρικές πρωταγωνίστρες, ως πολιτικοί και πολίτες. Ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα ως προς το κλίμα θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι για το παράδειγμα που δώσαμε. Η γυναίκα η οποία εμφανιζόταν ως ε, θύμα ε, στο, σε ζητήματα όπως η ανάπτυξη, η μετανάστευση, οι ε, καταστροφές τώρα εμφανίζεται με έναν ακόμα ρόλο θύμα αλλά και πρωταγωνιστής που δρά και που αγωνίζεται για αυτό που είναι πολύτιμο για τον πλανήτη. Υπάρχουν όμως επίγοντα θέματα. Στην έκθεση θελήσαμε να επιμείνουμε ότι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και πρέπει να καταστεί προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο προς την εξωτερική μας πολιτική όσο και την εσωτερική. Η ε, διακρίσεις που συνδέονται με την ισότητα των φύλων που είναι ε, παρούσες ε, στην κοινωνία μας και που συνδυάζονται και στις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή επιδεινώνονται. Άρα λοιπόν απαιτούνται ενέργειες για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Στην έκθεση αυτή ήθελα να περάσω τρία μηνύματα. Καταρχήν ότι είναι ευκαιρία η διάσταση της ισότητας των δύο φύλων. Με περισσότερη δικαιοσύνη και πιο αποτελεσματικά μπορούμε να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή ή να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Και θα πρέπει να δουλέψουμε ε, αντιμετωπίζοντας και την ανισότητα όσο και την κλιματική αλλαγή, δηλαδή οικονομική στήριξη και μέσα για την χειραφέτηση της, γυ... Ε, γυναίκας στην κοινωνία. Άρα λοιπόν αυτή η σχέση μεταξύ κλιματικής αλλαγής και χειραφέτησης γυναικών περνάει μέσα από μια διαδικασία ε, δικαιωμάτων και δεδομένων. Έτσι λοιπόν θα μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τη λήψη αποφάσεων όπως συνέβη με την πολιτική της ανάπτυξης τα τελευταία 20 χρόνια. Σε ολόκληρο τον κόσμο οι γυναίκες υφίστανται διακρίσεις επειδή είναι γυναίκες. Οι ανάγκες τους, οι επιδιώξεις τους, οι δυνατότητες είναι πολύ πιο περιορισμένες. Οι στατιστικές σε σχέση με την ισότητα των φύλων δείχνουν ότι υπάρχει διάκριση σε όλους τους τομείς της ζωής και σε όλες τις κοινωνίες. Έχουν λιγότερη πρόσβαση στην, στα χρηματοδοτικά μέσα, διαθέτουν λιγότερο το 1% των πόρων στον κόσμο, είναι το 70% των ατόμων που ζουν με λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα υποεκπροσωπούνται στη διαδικασία λήψης πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων, 19% ε, βουλευτές, 8% ως υπουργοί. Ε, ήδη τα είπαμε αυτά και εχθές, οι γυναίκες απασχολούνται ε, με δουλειά που δεν πληρώνεται, φροντίζοντας ε, παιδιά και ηλικιωμένα άτομα και τη δουλειά στο σπίτι και δουλεύουν σε παγκόσμιο επίπεδο για μόνο το 10% του παγκοσμίου εισοδήματος. Το 80% των μεταναστών ε, ενώ η θνησιμότητα είναι πέντε φορές μεγαλύτερη στο πλαίσιο των φυσικών καταστροφών. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχουν πολιτιστικά, οικονομικά, ε, νομικά και κοινωνικά εμπόδια ε, εις βάρος της γυναίκας και υπέρ των ανδρών. Και τούτο είναι εμφανές σε όλους τους τομείς οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό κλπ. Οι γυναίκες λοιπόν έχουν πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες προσαρμογής σε όλα τα θέματα που απαιτούν προσαρμογή στο πλαίσιο της αλλαγής του ε, κλίματος. Άρα λοιπόν αυτό, αυτή η τροτότητα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Έχει αναγνωριστεί ότι τούτο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής όλο και περισσότερα κείμενα όπως το ε, πλαίσιο για την καταπολέμηση των ε, φυσικών καταστροφών, η διακήρυξη του Ρίου του 1992 ε, λαμβάνουν υπόψη τις διακρίσεις βάρος των γυναικών σε όλες τις πτυχές της κλιματικής πολιτικής. Άρα λοιπόν η διάσταση της έλλειψης ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα επίγοντα και άμεσα προβλήματα όπως είναι οι φυσικές καταστροφές αλλά επίσης και να αντιμετωπίσουμε τα πιο μακροπρόθεσμα ε, προβλήματα της κλιματικής αλλαγής. Άρα λοιπόν ε, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη ανεξαρτησία και χειραγώγηση στις ε, γυναίκες. Τούτο σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει συμπληρωματικότητα ε, ε, ρόλων και επίσης είναι πολύ σημαντικό να αλλάξει η νοοτροπία που διαπερνά τις πολιτικές κλιματικής αλλαγής. Έτσι πρέπει να συμπεριληφθούν οι γυναίκες στις διαπραγματεύσεις αλλά και τους μηχανισμούς χρηματοδότησης με τη βελτίωση της παιδείας και της διαβούλευσης με τις γυναίκες και προωθώντας προγράμματα τα οποία δίνουν εξουσία στις γυναίκες στους κόλπους της κοινότητας όπου ζουν στις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά επίσης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά λοιπόν την συνειδητοποίηση όλων αυτών οι γυναίκες εν μέρη συμπεριλαμβάνονται. Έχει γίνει αυτή η διασύνδεση με μηχανισμούς αρρωγής και ανάπτυξης και ε, στις πολιτικές της αναπτυσσόμενες χώρες αλλά υπάρχει πλήρης απουσία στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά λοιπόν καθορίζονται οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την κατεύθυνση μιας πιο πράσινης οικονομίας και μιας προσέγγισης κατά τομής δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τη σχέση που, την διαφορά που υπάρχει μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ε, το ίδιο ισχύει και με τις πολιτικές της ενέργειας όπως έδειξε η έκθεση της κυρίας Εστρέλα εχθές ε, και στις μεταφορές και την γεωργία. Η καθοριστική τομή, λοιπόν για την μελλοντική ανάπτυξη της οικονομίας είναι κατά κύριο λόγο ε, συνδέονται κατά κύριο λόγο με την ανδρική παρουσία και δεν ευνοείται η ισότητα ανθρώπων και γυναικών. Διεύρυνση λοιπόν του οράματος έχει να κάνει με την δικαιοσύνη αλλά και με την αποτελεσματικότητα. Έτσι λοιπόν επιθυμούμε η σημασία της διάσταση της ισότητας των φύλων θα πρέπει να υπάρχει και να εμφανίζεται σε όλους τους τομείς και συνδέεται άμεσα με την εκπροσώπηση της γυναίκας, την πολιτική και την οικονομία. Η θέση σε ισχύ μιας πολιτικής υπέρ της ισότητας ανδρών και γυναικών απαιτεί καταπολέμηση των ανισοτήτων. Πολιτικές οι οποίες ε, διατυπώνονται χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την διάσταση της ισότητας κινδυνεύουν να καταλήξουν σε αρνητικά αποτελέσματα προς την ισότητα. Ε, η έλλειψη έρευνας στατιστικών στοιχείων σε τομείς όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, η ε, αγροτική πολιτική κλπ. είναι ε, η έλλειψη είναι εμφανής και απαιτούνται λοιπόν στοιχεία για να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Αυτά είχα να πω σχετικά με την έκθεση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές και εισηγήτρες για τις ιδέες που διατύπωσαν και είμαι στη διάθεσή σας να συζητήσω το περιεχόμενο και να έχουμε μια καρποφόρα συνεργασία ε, σχετικά με το θέμα αυτό στο πλαίσιο των θεσμικών μας οργάνων υπέρ των ε, συμπολιτών μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κιλ Νίλσεν. Ο λόγος της υπόλοιπης, η κυρία Στρέλα καταρχήν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας την κυρία Κιλ Νίλσεν. Η έκθεση της είναι καλά διατρομένη, πολύ ενδιαφέρουσα και βασίζεται, λαμβάνει υπόψη όλα τα, όλες τις τελευταίες εξελίξεις του Ντέρμπαν όπου οι γυναίκες ανέλαβαν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής ε, δεν ήταν τα αναμενόμενα βέβαια, αλλά ήταν θετικά και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην συμμετοχή των γυναικών. Η λίγη πρόοδος που έγινε μπορούμε να πούμε ότι οφείλεται στην αποφασιστικότητα που έδειξαν οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του Κλίματος. Χτες συζητήσαμε την έκθεσή μου για την ενεργειακή απόδοση και αυτά τα δύο θέματα συνδέονται μεταξύ τους ε, πολύ στενά. Και καθίσταται σαφές ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να αποκλειστούν από κανένα τομέα είτε της πολιτικής είτε της οικονομίας. Όπου υπάρχει ζωή εκεί πρέπει να είναι παρούσες και οι γυναίκες. Όπου λαμβάνονται αποφάσεις, εκεί πρέπει να συμμετέχουν και οι γυναίκες. Συμφωνώ με τις βασικές γραμμές της έκθεσης. Πιο συγκεκριμένα για το γεγονός ότι οι κλιματικές αλλαγές δεν είναι ουδέτερες σε ό,τι αφορά το φύλλο. Και αυτές οι αλλαγές έχουν διαφορετικές επιπτώσεις στο κάθε φύλλο είναι πολύ πιθανό να οξύνουν διαφορές που ήδη υπάρχουν ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών θα γίνουν πιο ε, σαφείς στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές του κόσμου. Το λέει και η έκθεση. Οι γυναίκες είναι πιο ευπαθείς στις κλιματικές αλλαγές και στις θεομηνίες δεδομένου ότι είναι θύματα πολλαπλών διακρίσεων, οι γυναίκες πλήττονται ιδιαίτερως επίσης από τη φτώχεια. Από την έλλειψη, η έλλειψη νερού και η ξηρασία αναγκάζουν τις γυναίκες να δουλεύουν περισσότερο για να εξασφαλίσουν τροφή, ενέργεια και νερό. Και πολύ συχνά οι νέες εγκαταλείπουν τη σχολική τους εκπαίδευση για να βοηθήσουν τις μητέρες τους σε αυτά τους τα καθήκοντα. Επίσης αξίζει να υποστηρίξουμε το ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε πλήρη συμμετοχή των γυναικών σε όλες τις πτυχές καταπολέμησης των, της κλιματικής αλλαγής. Οι γυναίκες θα πρέπει να είναι παράγοντες αλλαγής και η συμμετοχή τους στις κορυφή του κλίματος είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Οι γυναίκες θα πρέπει να συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με την καταπολέμηση και την προσαρμογή στην, στην ε, κλιματική αλλαγή σε όλα τα επίπεδα συμπεριλαμβανομένης και της έρευνας. Είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε την ανάγκη συμμετοχή των γυναικών στην έρευνα. Απ' την άλλη μεριά, δεδομένων των ευθυνών τους σε ό,τι αφορά την ε, διατήρηση σπάνιων ε, φυσικών πόρων οι γυναίκες θα έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην κλιματική βιωσιμότητα. Οι γυναίκες είναι ήδη πιο ευαισθητοποιημένες από τους άντρες σε ό,τι αφορά την βιωσιμότητα των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. Αυτή, η συνειδητοποίηση θα πρέπει, αυτή τη συνειδητοποίηση θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Του του λεχθέντος. Ως και την θα υποβάλω ε, ορισμένες τροπολογίες, ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ιδιαιτερότητα της φύσης των γυναικών σε θέματα όπως η ε, μετανάστευση και οι θεομηνίες. Θέλουμε, θέλω επίσης να τονίσουμε την ανάγκη της ένταξης του φύλου στην, στις αναπτυξιακές πολιτικές όπως για παράδειγμα στους στόχους χιλιετίας. Θα πρέπει η διάσταση του φύλου να ενταχθεί περισσότερο στην ε, ε, αναπτυξιακή μας πολιτική. Τελειώνω συγχαίροντας ξανά την εισηγήτρια. Η έκθεση είναι πολύ καλή και πιστεύω ότι θα συνεισφέρει έτσι ώστε ε, να ενισχύσουμε το ρόλο της γυναίκας της ε, σύγχρονης κοινωνίας και την μάχη ε, εν ώψη των προκλήσεων του μέλλοντος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Πιετικάινεν. Thank Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν και εγώ θα συγχαρώ την εισηγήτρια για την εξαιρετική της δουλειά σε αυτήν την έκθεση. Νομίζω ότι δίνει έμφαση στα κρίσιμα σημεία και στην δυναμική ε, πίσω από την κλιματική αλλαγή. Η, αναφέρει ότι οι γυναίκες είναι η πιο ευπαθής ομάδα και από οικονομικής πλευράς, αλλά και ε, ε, εξαιτία της γεωγραφικής κατανομής τους, όταν για παράδειγμα βρίσκονται σε χώρες που πλήττονται από έλλειψη φυσικών πόρων. Ε, πράγματι πλήττονται περισσότερο από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Είναι αλήθεια άλλωστε ότι οι γυναίκες δεν συμμετέχουν επαρκώς στη λήψη των αποφάσεων και δεν έχουν ε, πολιτική ισχύ και αυτό είναι ένα από τα σημαντικά προβλήματα. Υποστηρίζω λοιπόν πλήρως τις ιδέες που αναφέρει η έκθεση ότι ε, θα πρέπει να δώσουμε εξουσία στις γυναίκες στην πολιτική και σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή και σε, γενικότερα. Ε, κατόπιν ε, θα πρέπει στα συντάγματα μας να εντάξουμε το δικαίωμα σε ένα καθαρό περιβάλλον και το δικαίωμα στην πρόσβαση στους πόρους, στους φυσικούς πόρους εννοώ. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα βοηθήσει τις γυναίκες. Κατόπιν, αναφέρθηκε το θέμα των, της, των, των διακρίσεων στην πολιτική. Οι γυναίκες έχουν θέσεις στο περιβάλλον, την ε, εκπαίδευση ε, όταν έχουν κάποια εξουσία. Οπότε ε, αυτές οι γυναίκες που έχουν εξουσία, οι λίγες, έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τα πράγματα και πρέπει να το προσπαθήσουν. Χρειαζόμαστε όμως με περισσότερη συμμετοχή των γυναικών στη λήψη οικονομικών αποφάσεων. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω περισσότερο στην έκθεση το εξής. Την ε, ιδέα της θετικής εξουσίας, θετικής ισχύω. Ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός είναι γυναίκες. Οι γυναίκες είναι η πιο δραστήρια ομάδα στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και στην κοινωνία των πολιτών. Οι γυναίκες είναι αυτές που κυρίως μορφώνουν τα παιδιά. Οι Γυναίκες είναι αυτές οι οποίες ε, παίρνουν πολύ συχνά ε, τις καθημερινές αποφάσεις κατανάλωσης και συμμετέχουν πάρα πολύ στη λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο. Οπότε πιστεύω ότι θα έπρεπε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να δούμε πώς θα μπορούσαμε να στηρίξουμε περισσότερο τη συνεργασία, την οργάνωση, την αυτοοργάνωση και τις δραστηριότητες των γυναικών ω καταναλώτριες, ε, ω εκπαιδεύτριε και ο, ως άτομα που λαμβάνουν αποφάσεις σε τοπικό επίπεδο, γιατί εκεί θα μπορούσε να ξεκινήσει η αλλαγή πιο εύκολα. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ πολύ. Ε, και εγώ είχα εγγραφεί στον κατάλογο των ε, ομιλητών, μια και είμαι και σκιώδης εισηγητής θα ήθελα να πω ότι με βρίσκει απολύτω σύμφωνο ε, η άποψη της ε, συναδέλφου, ε, δηλαδή αυτά που ανέφερε η συγγήτρια είναι πάρα πολύ σωστά, καταδεικνύει σωστά το πρόβλημα και νομίζω ότι η σχέση κλιματικής αλλαγής και ε, ισότητας φύλων θα πρέπει να καταδειχθεί γιατί βεβαίως ε, η κλιματική αλλαγή επιδρά τα μάλα επί των γυναικών και θα πρέπει να αποσαφινιστεί ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζει τις γυναίκες η κλιματική αλλαγή και εδώ πραγματικά η συγγήτρια έχει αναφέρει όλα τα ε, ε, ουσιοδέστερα σημεία. Εγώ να προσθέσω μόνο δύο-τρία μικροπράγματα. Πρώτον, ε, θα πρέπει να εξηγήσουμε την, ε, τον, την αιτία, τον λόγο για τον οποίο ασχολούμαστε ε, με το θέμα αυτό. Ε, μιλάμε δηλαδή στην ουσία για την κατανάλωση, μιλάμε για τις καταναλωτικές συνήθειες των ανθρώπων, οι οποίοι ας πούμε καταναλώνουν πολλή ενέργεια, καταναλώνουν περισσότερο κρέας, ε, υπάρχουν κάποιες συνήθειες και κάποιοι καταναλωτικοί τρόποι ε, που θα πρέπει ε, να αναφερθούν γιατί επηρεάζουν την οργάνωση των πραγμάτων. Επίσης όσον αφορά αυτά τα στοιχεία α, β, γ, δ που συνδέονται με το σημείο 9 όπου ακριβώς υπογραμμίζεται η σημασία της γνώσης των γυναικών. Εγώ μπορώ να σας πω ότι ε, οπουδήποτε βελτιώθηκε η κατάρτιση των γυναικών είχαμε μια γενικότερη βελτίωση ε, ας πούμε ε, όσον αφορά την απερίμωση πληροφορώντας τις γυναίκες για το θέμα αυτό κερδίσαμε πολύ το ίδιο όσον αφορά την ενίσχυση της βιοπικιλότητας το ίδιο για την υπερθέρμανση Επομένως, ε, εάν ε, ε, σε περιοχές ας πούμε όπου οι γυναίκες έμαθαν πόσο βελτιώνεται η κατάσταση εάν φυτέψουν δέντρα, το έκαναν. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό οι γυναίκες να έχουν γνώσεις. Και ξέρουμε περιπτώσεις που οι γυναίκες έμαθαν να προβλέπουν στην ουσία καταστροφές ε, γιατί έμαθαν να διαβάζουν τα πρόδρομα σημάδια ε, και αποφεύθηκαν φυσικές καταστροφές ή μάλλον ε, θάνατοι λόγω των φυσικών καταστροφών. Άρα η γνώση των γυναικών είναι πάρα πολύ σημαντική. Όσον αφορά τώρα το τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από την πλευρά της Ευρώπης, μπορούμε να προκαλέσουμε κατά κάποιο τρόπο ε, τις ε, χώρες μας να καταρτιστούν ε, στόχοι όσον αφορά τα δικαστήρια. θα τα γράψω όλα αυτά, μην ανησυχείτε, θα τα καταλάβετε πολύ καλύτερα όταν θα τα δείτε γραμμένα. Αλλά πάντως είναι εξαιρετικής ποιότητας η έκθεσή σας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Άψογα, η κυρία Παπαδοπούλου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να πω ότι είναι μια πολύ ισορροπημένη έκθεση. Καταγράφονται όλα όσα πρέπει να αναφερθούν. Θα δώσω μια ιδιαίτερη βαρύτητα στη διάσταση των κλιματικών προσφύγων. Επειδή οι θεομηνίες επηρεάζουν πολλές περιοχές του πλανήτη και ιδίως αναπτυσσόμενες χώρες, όταν υπάρχουν ε, μεγάλες κλιματικές ε, ε, καταστροφές που οφείλονται στο στο κλίμα ε, βλέπουμε ότι ε, πολλοί κόσμοι, άνδρες και γυναίκες αλλά και παιδιά αναγκάζονται να αλλάξουν ε, χώρο όπου διαμένουν. Και εκεί ακριβώς βλέπουμε σε όλων των μεγαλείων τι σημαίνει κλιματικός πρόσφυγας και το βάρος πέφτει στους ώμους κυρίως των γυναικών όταν έχουν μικρά παιδιά, όταν έχουν μέλη ανάπηρα στην οικογένεια, όταν έχουν ηλικιωμένους τους οποίους φροντίζουν κυρίως οι γυναίκες και αντιλαμβανόμαστε όλοι όταν η ίδια οικογένεια χάνει την δική της οικογενειακή συνοχή και η οικογένεια είναι βασικό κύτταρο κάθε κοινωνία, οπωσδήποτε ε, κατά συνέπεια κινδυνεύει και η κοινωνική συνοχή. Επομένω, ε, εγώ προσωπικά θα ήθελα να ενισχυθεί ε, η μικροχρηματοδότηση σε γυναίκες, δηλαδή τα microloans τα οποία δίνονται, ούτως ώστε μετά οι γυναίκες να μπορέσουν να επαναδραστηριοποιηθούν οικονομικά μετά από τέτοιου είδους σαρωτικές αλλαγές στη ζωή τους, να μπορέσουν να έχουν κάποιους σπόρους ε, και μιλώ πάντα για τις αναπτυσσόμενες χώρες, ε, για να μπορούν να έχουν περισσότερες δυνατότητες διότι έχουμε δει από παλαιότερες εκθέσεις και του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών ότι όπου οι γυναίκες έχουν αναλάβει projects, προγράμματα μικροχρηματοδότησης τα λεφτά τα οποία εισπράττουν τα δίνουν για τα μέλη της οικογένειας και ιδίω για τα παιδιά και επομένως βοηθά κλιματικούς πρόσφυγες εάν στηρίζουμε τις γυναίκες οικονομικά να επαναδραστροποιηθούν για να μπορούν μετά να στηρίξουν τα μέλη της Είναι μια ψυχή στην οποία ε, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα γιατί είναι ένας πρακτικός τρόπος στήριξης των γυναικών. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ πολύ. Δεν ε, βλέπω κάποιον άλλον. Ε, να ζητάει τον λόγο. Μήπως ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελε να μιλήσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και καλημέρα σε όλους σας. Εξ ονόματος της Επιτροπής και την αρμόδια Γενική Διεύθυνση για το κλίμα θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ε, έκθεση αυτή. Όπως υπόθηκε και προηγουμένως, είναι γεγονός ότι στην ευρύτερη συζήτηση για την κλιματική αλλαγή παραμερίστηκε, παραγκονίστηκε συχνά το θέμα των ε, γυναικών. Ε, είναι σαφές ότι θα πρέπει να ε, έχουμε όλο και, περισσό, πιο φιλόδοξους στόχους για το 2020, δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στις αναδυόμενες οικονομίες, αναπτυσσόμενες χώρες. Και ε, βεβαίως είναι γεγονός ότι οι γυναίκες στις ε, λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και στις πιο φτωχές χώρες είναι αυτές ε, οι οποίες θα πληγούν περισσότερο από τις κλιματικές αλλαγές. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει άμεσα να σταματήσουν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Είναι γεγονός επίσης ότι θα πρέπει όσον αφορά τον καταμερισμό εργασίας, όσον αφορά ε, τη θέση των ανδρών και των γυναικών στην κοινωνία, να κατανοήσουμε ε, την έλλειψη ισορροπίας και ισοτιμίας ε, και επομένως να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα. Οι στόχοι που αναφέρονται εδώ βρίσκουν σύμφωνοι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. λαμβάνουμε ε, μέτρα τα οποία αφορούν συγκεκριμένα την αντιμετώπιση της ισότητας των φύλων ε, και απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Επίσης ε, θεωρούμε ότι η ισότητα των φύλων είναι σημαντικό στοιχείο της αναπτυξιακής πολιτικής ε, και για το 2015 και 2020 για τους στόχους αυτούς ε, ε, οι γυναίκες παίζουν σημαντικό ρόλο. Στο πρόγραμμα στη χρονική περίοδο 2010-2015 όσον αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία επίσης οι γυναίκες παίζουν σημαντικό στο τέλος του 2012 το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων θα έχει ε, καθορίσει και τις αρμοδιότητες ε, του ε, Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων και θα δοθεί και η τελική μορφή των δικτών ε, που θα αποφαίνονται για την ε, επιρροή ε, της κλιματικής αλλαγής στις γυναίκες και στην ισότητα των φύλων γενικότερα. Θεωρούμε ότι και για τη στρατηγική 2013 η θέση των γυναικών είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, και ε, το Νοέμβριο ε, είχε έρθει η Επίτροπος η οποία είναι αρμόδια για τα θέματα αυτά στην Επιτροπή σας και αναφέρθηκε για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε να, με τον οποίο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της θέσης των γυναικών στις λιγότερο, στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει γνώση όλων των ετοιμάτων που έχουν υποβληθεί μέσω της της εκθέσεως ημερίζεται τους στόχους και βεβαίως θα αξιολογήσει τους στόχους αυτούς σε ευθέτω χρόνο ε, και θα επανακάμψουμε ε, αναφέροντας ότι μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κιλνένσεν για να ολοκληρώσει. Ε, ναι, χαίρομαι βεβαίω γιατί φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν πολλέ τροπολογίε οι οποίε βεβαίω θα βελτιώσουν την έκθεση και επομένω ε, περιμένω τι τροπολογίε σα. Αυτό ήθελα να πω μόνο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Κλείνει λοιπόν και αυτό το σημείο. Θα ήθελα να σας ε, ξεκαθαρίσω το χρονοδιάγραμμα. Τροπολογίες, ε, προθεσμία υποβολής τροπολογιών 10 Ιανουαρίου. Θα το συζητήσουμε στις 25-26. Θα ψηφίσουμε 27-28 Φεβρουαρίου και θα έρθει στην Ολομέλεια του Μαρτίου ή του Απριλίου. Και τώρα επανερχόμαστε ε, μάλλον ερχόμαστε στο σημείο 14 γυναίκες στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων ποιότητα και ισότητα και δίνω το λόγο στην κυρία Πιέτη Κάινεν. Ε, poliittisena päätöksentekijöinä on kysymys sekä laadusta että tasa-arvosta. Tasa-arvosta ε, έχει μεγάλη σημασία η ποιότητα αλλά και η ισότητα, διότι οι άνδρες και γυναίκες έχουν τα ίδια δικαιώματα ε, σύμφωνα με την ε, χάρτα και έχουν ίσα δικαιώματα στην προετοιμασία και την εκπόνηση. Ισότητα λοιπόν γιατί, γιατί οι γυναίκες ανήκουν στην ομάδα εκείνη που εξαιρείται, που απέχει περισσότερο ε, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ταυτόχρονα είναι και θέμα ποιότητας. Γιατί, διότι όσο περισσότερο η δομή της λήψης αποφάσεων αποκτά ποικιλία, τόσο περισσότερο αντιπροσωπευτική της πραγματικότητας καθίσταται. Αυτή τη στιγμή αυτό που μας απασχολεί στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το γεγονός ότι ε, η εξέλιξη προς την συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα είτε καθυστερεί είτε αναστέλλεται. Υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Ε, δηλαδή θα θέλαμε πάρα πολύ να ε, υπάρχει μια κατανομή 50-50 ή 60-40. Ωστόσο, ποια είναι ε, τα προσκόμματα ή οι φραγμοί που εγείρονται. Υπάρχουν ε, διαρθρωτικά ε, προβλήματα, παραδείγματος χάρη κενά ή ελλείψεις όσον αφορά τη δομή, τις κρατικές δομές την ε, μέρημνα των ε, παιδιών, των ηλικιωμένων. Η οικονομική και κοινωνική κατάσταση των γυναικών είναι ε, χειρότερη. Υπάρχουν λοιπόν συνθήκες, συνθήκες οι οποίες εμποδίζουν τις γυναίκες να συμμετάσχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να αναλάβουν την ευθύνη για το μέλλον της κοινωνίας. Από την άλλη υπάρχουν πολύ ισχυρά, δυνατά στερεότυπα στα μέσα ενημέρωσης, στις δομές λήψης αποφάσεων, στα κόμματα τα πολιτικά. που θέτουν, τοποθετούν τις γυναίκες μέσα σε ε, περιοριστικά όριο σε περιορισμούς, σε κουτιά θα μπορούσε κανείς να πει μεταφορικά. Δεν φταίνει οι γυναίκες ε, για την κατάσταση αυτή. Δεν είναι οι γυναίκες οι οποίες προτιμούν να ασχολούνται μόνο με τα παιδιά, αλλά υπάρχουν δομικά εμπόδια ή δομικοί λόγοι εξαιτία των οποίων οι γυναίκες δεν έχουν την ίδια δυνατότητα να συμμετάσχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Πέραν ε, τούτου, η ίδια η δομή της πολιτικής, των, των πολιτικών κομμάτων είναι διαφορετική όσον αφορά τις υποψήφιες γυναίκες. Πώς ε, οι μηχανισμοί των πολιτικών κομμάτων διευκολύνουν ή εμποδίζουν τη συμμετοχή των ε, γυναικών και πώς επίσης ε, η πολιτική εξουσία, η ισχύς εντός των κομμάτων ασκείται διακρίσεις εις βάρος των γυναικών ως προς την λειτουργία του κόμματος, την αποστολή της εξουσίας. Ε, όλα αυτά έχουν τις αρνητικές τους επιπτώσεις στην εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική. Η ανάληψη ευθυνών σε κοινωνικό επίπεδο, σε επίπεδο παιδείας, κατανομής ε, ενώ από την άλλη οι άνδρες είναι αυτοί οι οποίοι κρατούν στα χέρια τους την λήψη αποφάσεων στη χάραξη των βασικών ε, γραμμών πολιτικής. Σε οικονομικό επίπεδο επίσης οι γυναίκες βρίσκονται σε μειονεκτικότερη θέση. τα ε, ε, συστήματα, τα, μάλλον ε, στις δομές της εκστρατείας. Οι πόροι οι οποίοι διατίθενται υπέρ των ανδρών ή υπέρ των γυναικών, όταν γίνονται οι επιλογές, όταν οι υποψήφιες προστρέχουν στους πόρους που είναι διαθέσιμοι και εκεί υπάρχει διάκριση εις βάρος των γυναικών. Η γυναίκα λοιπόν ως πολιτικός που λαμβάνει αποφάσεις ε, εκπροσωπείται ελιπώς. Από την άλλη, όταν κατανέμονται οι αρμοδιότητες και οι υπευθυνότητες και πάλι υπάρχει μια ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, όλα αυτά γίνονται περισσότερο από τους άνδρες. Η προετοιμασία των επιτροπών, οι ε, ανώτεροι αξιωματούχοι οι οποίοι λαμβάνουν τις πολιτικές αποφάσεις. Στο επίπεδο αυτό πράγματι υπάρχει υποεκπροσώπηση των γυναικών και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Ζούμε σε μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία στην οποία απαιτείται πολλή προετοιμασία, υπάρχουν διαδικασίες και και ακριβώς και στο επίπεδο της προετοιμασίας όσο και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται. Και το βλέπει αυτό κανείς όταν ασκεί κάποιες αρμοδιότητες. Βλέπουμε τις γυναίκες να είναι πάρα πολύ δραστήριες ε, σε επίπεδο κοινωνίας πολιτών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Κύριε Πρόεδρε, στην έκθεση αυτή προσπάθησα να καταρτήσω έναν κατάλογο πολύ συγκεκριμένο και έναν κατάλογο εργαλείων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ώστε να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες που υπάρχουν, ώστε στο μέλλον να καταλήξουμε σε περισσότερη ισότητα. Προτάσεις σε επίπεδο εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό. Στρατηγικές που λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα κίνητρα και ελαττήρια διακρίσεων εις βάρος των γυναικών. Λείπουν λοιπόν δομές στο κράτος πρόνοιας, στο κράτος ευμερίας, η έλλειψη βασικών κοινωνικών υπηρεσιών στις οποίες ε, πρέπει να έχουν πρόσβαση οι γυναίκες, συνδυασμός οικογενειακής ζωής με επαγγελματική που εξαρτάται ακριβώς από αυτές τις δομές και που θα μπορέσει να βοηθήσει τις γυναίκες ε, βοήθεια στην, στην πολιτική ε, αρρωγή μάλλον των γυναικών ώστε να αναπτύξουν ε, ε, πολιτικές. Το ίδιο ισχύει για το εσωτερικό των κομμάτων, την κατάρτιση του καταλόγου των ε, υποψηφίων και την κατάληψη σημαντικών θέσεων στην ιεραρχία από τις γυναίκες. Προτροπή των κομμάτων να συμπεριλάβουν τις ε, γυναίκες, αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης των πολιτικών ε, κομμάτων, η ισότιμη ε, προσέγγιση ανδρών και γυναικών υποψηφίων ούτως ώστε να εκπροσωπούνται πολύ περισσότερο οι γυναίκες. Επίσης υπάρχουν κάποια θέματα σε σχέση με τις ποσοστώσεις, αυτά θα πρέπει να τα επανεξετάσουμε και να σκεφτούμε πάνω σε αυτό το θέμα των ποσοστώσεων. Οι ίδιες αρχές θα πρέπει να ισχύουν όταν οι χώρες μέλη προτείνουν υποψηφίους για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι πρέπει να, υπάρχει, να υπάρχουν δύο υποψήφιοι, άνδρες και γυναίκα, όπως επίσης και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη σύνθεση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει πάντα να υλοποιείται αυτός ο στόχος της ισότητας, της ίσης εκπροσώπησης των δύο φύλων. Επίσης, ε, στον διορισμό ε, υψηλόβαθμων αξιωματούχων και εκεί ε, ενδεχομένως πρέπει να εφαρμόζεται μια ποσόστοση σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως και σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, Ε, θα πρέπει να διατυπώσουμε την ευχή και την προτροπή προς τα εθνικά κοινοβούλια ώστε να λειτουργήσει αυτή η ίση εκπροσώπηση ε, τόσο ως προς τα μέλη όσο και στα προεδρία, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, πρόεδροι επιτροπών και καθ' όλη τη διάρκεια της εντολής μάλιστα για να μπορέσουμε να επιτύχουμε επιτέλους αυτό το στόχο του 50%. Ε, ενδεχομένως θα πρέπει να καθορίσουμε μια, ε, ένα χρονοδιάγραμμα ε, διάρκας ας πούμε τριών, εντο, τριών θητιών, τριών εντολών του Κοινοβουλίου. Η στρατηγική από μόνη της βεβαίως δεν αρκεί. Απαιτούνται έρευνες και καλύτερες έρευνες μάλιστα. Προγράμματα έρευνας, παρακολούθησης και επιθυμούμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαθέσει επαρκή κονδύλια για τις έρευνες αυτές για να γίνει μια καλύτερη αξιολόγηση από αυτήν που έχουμε μέχρι σήμερα. Απαιτούνται διαδικασίες και σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο για να δούμε ποιοι είναι οι λόγοι που εμποδίζουν, που προβάλλουν προσκόμματα στην επίτευξη των στόχων που θέτουμε, ώστε να αναλυφθούν μέτρα ξεκάθαρα για να επέλθει διόρθωση στις πολιτικές που ασκούνται. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί μου, τη γραμματεία, τους κοιόδης εισηγητές και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να δουλέψουμε καλά και πιστεύω ότι η εμπειρία που θα αποκομίσουμε θα είναι επικοδομητική. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα έχετε το λόγο για τη συζήτηση. θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγητρία για αυτή την πολύ καλή έκθεση Όλοι νομίζω συμφωνούμε πως η ποιότητα των αποφάσεων εξαρτάται από την ποιότητα αυτών που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Πιστεύω ήγη ότι οι γυναίκες δεν θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν μόνο το 10 ή το 20% αυτών που λαμβάνουν αποφάσεις, όσο το δυνατόν περισσότερους, όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν. Ακόμα και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακόμα και εδώ στην ομάδα μας και ε, πρέπει να συμβαίνει το αντίστοιχο, δηλαδή μεγαλύτερη συμμετοχή ανδρών στην ομάδα μας. Και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να εντάξουμε τους άντρες στις γυναικείες οργανώσεις. Οι περισσότερες κοινωνίες δεν παίρνουν στα σοβαρά το θέμα της ισότητας των δύο φύλων. Όμως ε, η αλλαγή ξεκινάει από τα ίδια τα μυαλά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βιλμπάου. Καταρχήν να συγχαρώ την εισηγήτρια για τις προσπάθειες της. Στις 3 το απόγευμα κλείνει η προθεσμή για την υποβολή τροπολογιών. Ε, εμείς θα υποβάλουμε μερικές υποστηρίζοντας το περιεχόμενο της έκθεσης. Είναι θέμα δικαιοσύνης αλλά κυρίως δημοκρατίας. Εμείς αντιπροσωπεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από το 50% του πληθυσμού. Συνεπώς θα πρέπει και η συμμετοχή μας να είναι ισότιμη και ισόρροπη. Ε, θα ήθελα απλώς να χρησιμοποιήσουμε ε, την ορολογία που χρησιμοποιούμε ως τώρα στα κείμενά μας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε διεθνή ε, κείμενα και σε κείμενα σε εθνικό επίπεδο. Οι τροπολογίες μας έχουν σχέση με συγκεκριμένα θέματα ε, σχετικά με τα πολιτικά κόμματα και τα συνδικάτα, συνδικάτα στα οποία δεν αναφέρεται η έκθεση καθόλου. Και τα συνδικάτα έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη συλλογική δράση, στους τόπους εργασίας, οπότε έχουν και ευθύνες θεσμικής φύσεως. Αυτό που βλέπουμε σε όλο τον κόσμο και επίση στην Ευρώπη, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ε, Έχουμε δει ότι ε, διοικητικά μέτρα έχουν βελτιώσει τη συμμετοχή των γυναικών. Συνεπώς, ξέρουμε ποια είναι τα μέτρα τα οποία είναι αποτελεσματικά. Και νομίζω ότι με τέτοιου είδου μέτρα μπορούμε να προχωρήσουμε. Λείπει από την έκθεση επίσης ένα από τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην συμμετοχή τους σε κοινοβουλευτικά καθήκοντα, που είναι το θέμα των αντικαταστάσεων. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν προβλέπει την αντικατάσταση των γυναικών σε κανένα από τα κοινοβούλια όταν, για παράδειγμα, ε, γεννήσουν ε, ένα παιδί κατά τη διάρκεια της ε, άδειας μητρότητάς του στο δικό μας κοινοβούλιο στην Ισπανία είχαμε τρομακτικά προβλήματα διότι είχαμε γυναίκες οι οποίες ήταν έτοιμες να γεννήσουν ε, και δεν μπορούσαν να χάσουν ε, ούτε τις ψηφοφορίες που λάμβαναν χώρα στο κοινοβούλιο διότι δεν μπορούσαν να αντικατασταθούν. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να προτείνουμε λοιπόν συγκεκριμένα μέτρα σε συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και που τις εμποδίζουν στην ομαλή συμμετοχή τους στην, στο πολιτικό πεδίο. Πρέπει να προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα έτσι ώστε να ε, αλλάξει, να τροποποιηθεί η ε, διοικητική νομοθεσία αλλά και η εκλογική νομοθεσία. Η εκλογική νομοθεσία η οποία περιλαμβάνει τους κανόνες για την υποβολή λίστας κάθε κόμματος. Οι λίστες θα πρέπει να είναι ισόρροπες έτσι ώστε να ε, προβλέπεται συμμετοχή των γυναικών σε επίπεδο 50% ενδεχομένως. Θα πρέπει οι κανόνες που θα θεσπιστούν να μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε το κατά πόσον εξασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών στη συμμετοχή τους στις εκλογές. Ε, είπα λοιπόν θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες. Ε, γιατί ε, δεν πρέπει να δράσουμε μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Η Ευρώπη είναι Ένωση Κρατών αλλά και Περιφερειών και οι Περιφέρειες έχουν πολλές καλές εμπειρίες. Το 2005 η χώρα των Βάσκων υιοθέτησε ένα νόμο για την ισότητα των δύο φύλων τροποποιώντας τις, ε, την εκλογική νομοθεσία και την ε, νομοθεσία περί κρατικών υπηρεσιών εις τρόπον ώστε να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών και στις δημόσιες υπηρεσίες, στον κρατικό τομέα και στο τοπικό κοινοβούλιο. Στην έκθεση επίσης υπάρχει κάτι το οποίο δεν είχα καταλάβει καλά και θα ζητήσω με τροπολογία. Σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση των γυναικών σε, ερετά, σε θέσεις, ε, ε, αναφέρεται σε ένα ποσοστό 50% για τρεις τουλάχιστον θητείες. Όχι, εγώ πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να είναι κάτι μόνιμο. Θέλουμε να καταργηθούν οι ποσοστώσεις, ε, ε, θέλουμε να μην περιοριστεί αυτή η ποσόστοση στις τρεις ε, θητείες. Ε, τέλος, στα μέτρα για την υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών, στο σημείο 16, κάνουμε λόγο στην ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και την εργασιακή ζωή και την κατανομή ε, του, του κόστους ε, πατρότητας ανάμεσα στους εργοδότες και τους εργαζόμενους. Δεν πρέπει να μιλήσουμε μόνο, μιλήσουμε μόνο για το κόστος πατρότητας, αλλά και μητρότητας. Νομίζω ότι και τα δύο είναι σημαντικά. Επίσης να υπενθυμίσουμε ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυσκολευόμαστε να πείσουμε τα κράτη-μέλη να δεχτούν ε, η αμοιβή του καινούριου πατέρα, νέου πατερινέας μητέρας κατά τη διάρκεια της ε, άδειας μητρότητας ή πατρότητας να είναι το 100%, στο 100% του μισθού. Επίσης, πρέπει να δούμε το, την εικόνα που δίνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. κοιτάξτε τις εφημερίδες τη σημερινή, τη χθεσινή, του προηγούμενου μήνα, ποια είναι η εικόνα της γυναίκας. Ε, που ε, εμφανίζεται είναι ανύπαρκτη κατά βάση. Και οι τίτλοι που συνοδεύουν πολύ συχνά τις, ε, τα άρθρα ε, και την εικόνα της γυναίκας δεν είναι πολύ θετικοί. Ε, συζητώντας ποια γυναίκα μπορεί να είναι σημαντική για την Ευρώπη, όλοι μας, ε, όλων μας το μυαλό πηγαίνει στη Μέρκελ. Αλλά η Μέρκελ είναι η μόνη γυναίκα τελικά που εμφανίζεται συχνά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ποιες είναι οι υπόλοιπε γυναίκες, ελάχιστες. Αν πάρουμε την έκθεση, μια οποιαδήποτε έκθεση, έκθεση των ΗΕ για παράδειγμα, ε, θα δούμε ότι η παρουσία των γυναικών στην λήψη των αποφάσεων ε, συνεισφέρει την κοινωνική ευημερία, στην ευημερία των παιδιών, στην αλληλεγγύη, στη μείωση της διαφθοράς, ε, στην πιο αποτελεσματική διαχείριση και Τέλο να πω ότι η εικόνα των ανδρών στα, σε διεθνές επίπεδο ε, συνδέεται με τη συγκρούση, ενώ η εικόνα των γυναικών με την ειρήνη. Ε, να αναφερθώ στις γυναίκες με τα μαύρα, στις γυναίκες με τα λευκά. Οι γυναίκες πάντοτε συνδέονται με προσπάθειες ειρήνευσης. Συνήθως έχουμε πολλούς ε, λόγους για να ε, εργαστούμε επί της ενίσχυσης του ρόλου των γυναικών στη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Ευχαριστώ. Tack för det och då går ordet till... Ευχαριστώ. Η κυρία Παπαδοπούλου. Thank you. I also Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια κυρία Πέτη Κάνεν ε, για την πολύ καλογραμμένη έκθεσή της που υπογραμμίζει την ανάγκη για ποσοστοποιημένους στόχους ε, διαρκείς μηχανισμούς ε, εποπτείας. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολλά εργαλεία τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και πρέπει να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε ε, να καλυφθεί ε, το χάσμα ανάμεσα στην ομοθεσία και την πραγματική ζωή. Είμαι ε, σκιώδης συγγήτρια των σοσιαλιστών και δημοκρατών και είναι γεγονός ότι υποεκπροσωπείται η γυναίκα και στις, στο δημόσιο διοίκηση και στην οικονομική διοίκηση και στην εξωτερική πολιτική αλλά και αλλού πρέπει να αναλαμβάνουν ηγετικέ θέσεις ε, και βλέπουμε ότι ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μονάχα το 1 τρίτο ε, των υψηλόβαθμων υπαλλήλων είναι γυναίκε και μάλιστα δεν έχει αλλάξει το στοιχείο αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι γεγονός ότι η έκθεση έχει όλα τα στοιχεία τα οποία πρέπει να αναφέρουμε, το ρόλο των μέσων ενημέρωσης, των πολιτικών ομάδων, των πολιτικών ε, κομμάτων, ε, το, της, ε, των κυβερνήσεων, αλλά Πιστεύω ότι εάν τα μέτρα γίνουν ε, νομικώς δεσμευτικά όσον αφορά ε, τις ε, ποσοστώσεις για εκλόγιμες θέσεις, αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Από την άλλη πλευρά βέβαια, κάθε πολιτικό κόμμα έχει διαφορετικό τρόπο ορισμού των υποψηφίων και οι γυναίκες οπωσδήποτε στην κατάρτιση των πολιτικών ε, ληστών δεν έχουν ε, το ίδιο βάρος ε, και την ίδια πρόσβαση με τους άντρες. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπογραμμίσουμε την ανάγκη τα εργαλεία αυτά να είναι δεσμευτικά, την ανάγκη να ληφθούν νομικά μέτρα και βεβαίως να είναι υποχρεωτικά και τα συστήματα των ποσοστώσεων καθώς επίσης να υπάρξουν και εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Τελευταίο μου σχόλιο. Υπάρχουν υπερβολικά πολλά ψηφίσματα για το θέμα αυτό ε, και από πολλά διεθνή σώματα. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα, η Πλατφόρμα της Νέας Υόρκης, ε, ψηφίσματα από το, ε, από το Συμβούλιο της Ευρώπης, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό που χρειαζόμαστε στην ουσία είναι ε, μια καλή πρακτική που θα απομονώσουμε σε κάποια χώρα και ξέρουμε ότι στις σκανδιναβικές χώρες οι πρακτικές ε, ε, ενθάρρυνσης συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική ζωή είναι καλές. Και έχοντας αυτές τις καλές πρακτικές από μια χώρα να προσπαθήσουμε να τις εφαρμόσουμε στις άλλες χώρες. Γιατί διαφορετικά εάν κάθε χώρα μέλος αποφασίζει μόνη της για τον τρόπο με τον οποίο θα επιδιώξει και θα επιτύχει εν τέλει την ισότητα θα χάσουμε πολύ χρόνο. Να δούμε σε ποιε χώρε κάποια εργαλεία, κάποια μέσα είναι πιο αποτελεσματικά και να το εφαρμόσουμε και στι άλλε χώρε. Ε, κατά αυτή την έννοια λοιπόν θα υποβάλουμε και τις ε, τροπολογίε μα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ έχω εγγραφεί στον κατάλογο των αγορητών. Είμαι σκιώδης εισηγητής. και νομίζω όπως και η ίδια η και ε, οι σκιώδες που πήραν το λόγο ότι στην έκθεση αυτή πραγματικά με πολύ σαφήνεια ε, περιλάβαμε όλα τα στοιχεία τα οποία πρέπει να αναφερθούν. Ε, ε, η δουλειά είναι πάρα πολύ καλή, γίνεται λόγος για πράξεις και όχι για λόγια ε, και πραγματικά είναι πολύ σημαντικές οι προτάσεις προς την κατεύθυνση της διαφάνειας και της αφήνειας. Δεν έχω πολλές τροπολογίες, μερικές τροπολογίες μονάχα. γίνεται πολλής λόγος ε, για τις ε, ποσοστώσεις. Η άποψή μου όμως είναι ότι σε φυσιολογικές συνθήκες εξετάζοντας ε, την ε, κατανομή ε, των θέσεων θα πρέπει να βασιστούμε στις γνώσεις και την αξία το να πούμε 50% γυναίκες και 50 άνδρες αυτό θα, θα ήταν το φυσιολογικό εάν δεν φτάσουμε σε αυτό το φυσιολογικό αποτέλεσμα σημαίνει ότι ένα τμήμα του πληθυσμού δεν είχε πρόσβαση στη σωστή γνώση ε, είναι γεγονός ότι οι άνδρες συνήθως επιλέγουν άνδρες ή ενθαρρύνουν άνδρες. Ε, τα αγόρια μεγαλώνουν ε, σε ένα περιβάλλον, περιβάλλον όπου τους τονίζουν τα χαρακτηριστικά τους θα πρέπει να ληφθεί υπόψη επομένως και η κοινωνική διάσταση της κοινωνίας μας έτσι όπως είναι οργανωμένη τώρα. Νομίζω πάντως ότι θα πρέπει να σχηματοποιηθούν οι ποσοστώσεις να γίνουν πιο συγκεκριμένες. Επίσης, σε κάποια σημεία της έκθεσης θα μπορούσαμε ίσως να γίνουμε πιο ισχυροί, πιο δυνατοί, στο σημείο 3 ας πούμε, που το Κοινοβούλιο κάνει έκκληση στις χώρες Ε, νομίζω ότι εδώ μπορούμε να γίνουμε λίγο πιο ισχυροί και όπως λέει και η κυρία Μπιλμπάου ε, αυτές ε, οι τρεις ε, θητείες ε, είναι ένα σημείο σημαντικό. Στο σημείο 9 επίσης ε, το Κοινοβούλιο καλεί το Συμβούλιο και την Κομισιόν να υπογραμμίσει, να βελτιώσει την ισότητα όπου δει, όπου δει παντού χρειάζεται. Ε, δηλαδή αυτό καταλαβαίνετε πολύ μικρές ε, προσθήκες και μικρές ε, τροποποιήσεις όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις επίσης νομίζω ότι όταν ε, στέλνουμε τις αντιπροσωπείες μας σε εξωτερικές αποστολές, ναι, πρέπει να δούμε τη σύνθεση των αποστολών. Ε, ίσως είναι δύσκολο να πούμε ότι πρέπει να το κάνουμε, αλλά πάντως να λαμβάνεται υπόψη η ισότητα των φύλων όταν αποφασίζουμε ποιος θα συμμετάσχει σε κάποια αποστολή. Γιατί να στείλουμε με δύο άντρε στην Κοπενχάγη, μπορεί να πάει μια γυναίκα και ένα άντρα. Ε, Στι αντιπροσωπείε λοιπόν να υπόψη το θέμα ε, τη ισότητα των φύλων. Επίσης, αν ε, ως εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν συναντιόμαστε με τρίτες χώρες, με εκπροσώπους χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να δείξουμε μια καλή εικόνα και δεν μπορεί να πάω εγώ μόνος μου ας πούμε σαν πρόεδρος θα πρέπει να υπάρχει και κάποια γυναίκα η οποία θα μιλάει ε, ε, εξ ονόματος ε, της Επιτροπής γιατί συχνά βλέπουμε ότι στις συνεδριάσεις μόνο οι άντρες παίρνουν το λόγο ας πούμε. Και νομίζω ότι και στα briefing notes θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε και το, η διάσταση του φίλου. Πάντως, η έκθεση είναι πάρα πολύ καλή, είναι σαφής και σε ευχαριστούμε για την έκθεση αυτή. Κύριε Κιλ Νίλσεν, να επανέλθω σε ένα σημείο το οποίο σχολιάστηκε, το θέμα των πολιτικών κομμάτων και το πώς μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο. Είμαι υπέρ της ανάγκης δεσμευτικών νομικών μέτρων. Όχι εξαιτία μιας ιδεολογίας, αλλά λόγω της εμπειρίας μου. Στην Γαλλία ανήκω σε ένα πολιτικό κόμμα, τους πράσινους, που στο καταστατικό μας έχουμε γράψει την ισότητα, έχουμε γράψει την ισότητα το 1984 ήδη ισότητα και σε ό,τι αφορά την εσωτερική μας οργάνωση και σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στις λίστες. Και αυτό έδωσε αποτέλεσμα γιατί ήμασταν η πρώτη στη Γαλλία που είχαμε γυναίκα πρόεδρο περιφέρειας, είχαμε γυναίκα υποψήφια για την Προεδρία της Δημοκρατίας στη Γαλλία και τώρα θα έχουμε μία. Ε, έχουμε επίσης ε, οκτώ γυναίκες στους, μεταξύ των 14 που ε, μας εκπροσωπούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το γεγονός ότι εγγράψαμε λοιπόν στο καταστατικό μας ε, την ισότητα μας την υπέβαλε και αυτό έδωσε αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να γίνει και αλλού. Το έχω ζήσει, είμαι πεπισμένη γι' αυτό. Στην παράγραφο 3 λοιπόν, να μην πούμε όταν αυτό είναι δυνατό. Πρέπει να το διαγράψουμε αυτό. Πρέπει να την απαιτήσουμε την ισότητα. Η ποσόστοση ω όρο δεν, μου αρέσει. Θα πρέπει να μιλάμε για ισότητα ή ισότιμη συμμετοχή, ίση συμμετοχή. Ε, όχι ποσόστοση. Οι ποσοστώσει είναι ποσοστά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλου τύπου πράγματα και αντικείμενα. Για παράδειγμα, ε, επαγγελματική ε, ε, ε, συμμετοχή κατά επάγγελμα, τόσα τα εκατό αγρότες, τόσα τα εκατό εκπαιδευτικοί κλπ. Εδώ μιλάμε για ισότητα, για ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών. Ευχαριστώ. Eh, πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ. Η Κομισιόν. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de me donner euh, la parole. En effet, euh, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται για μια έκθεση πολύ σημαντική, διότι έχει να κάνει με την ε, μη επαρκή εκπροσώπηση των γυναικών σε επίπεδο λήψης αποφάσεων. Αυτή η ανησυχία ε, περιλαμβάνεται και σε έναν από τους πέντε βασικούς τομείς της δράσης και της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα ισότητας ανθρώπων και γυναικών για την περίοδο 2010-2015. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την πρόθεση να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των γυναικών στις προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με προγράμματα χρηματοδότησης, ε, προγράμματα στο πλαίσιο των θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, και της ε, ηθαγένειας Ευρώπη υπέρ των πολιτών. Η Κομισιόν υποστηρίζει την έννοια που μάλλον το στοιχείο που τονίζει η έκθεση ότι είμαστε υπέρ της βάσης δεδομένων που δημιουργήθηκε το 2004 που μας δίνει ε, στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ε, ζωή τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε εθνικό αλλά επίσης και στην οικονομική και την διοικητική ζωή αλλά και στο δικαστικό τομέα. Η Κομισιόν επιθυμεί να ευχαριστήσει για την υποστήριξη προς την ε, πρωτοβουλία αυτή μέσω της έκθεσης. Όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις, τις οποίες ε, θίγει το σχέδιο έκθεσης, η ε, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης καταβάλει προσπάθεια ώστε να βελτιωθεί η εκπροσώπηση των γυναικών στον τομέα δραστηριοτήτων της, τόσο ως προς την εκπροσώπηση όσο και στην εξωτερική πολιτική. Δεν θα αναφέρω όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί, αλλά να αναφέρω ενδεικτικά ότι δημιουργήθηκε το UN Women, ο ΙΕ γυναίκες, ε, ιδρύθηκε φέτος, η ε, Κομισιόν δεσμεύθηκε να συνεργαστεί πολύ στενά με αυτό το νέο φορέα του ΟΗΕ για να υπάρξει μια στρατηγική εταιρική σχέση και να έχουμε ε, πιο απτά αποτελέσματα στον τομέα της ισότητας ανδρών και γυναικών. Υπάρχει και ένα μνημόνιο συναντήληψης που δίνει το πλαίσιο αυτής της ετελικής σχέσης ε, βρίσκεται στη φάση της εκπόνησης. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εποπτεία επιτήρηση των εκλογών. Εκεί αναπτύσσονται σχέσεις όπου θα πρέπει να περιλαμβάνεται αυτή η διάσταση της ισότητας των ε, γυναικών με τους άνδρες τόσο ως προς την, ε, τον, τους υποψηφίους όσο και τον έλεγχο, την εποπτεία των εκλογών. Έτσι λοιπόν, οι γυναίκες ως πρωταγωνιστές στην οικοδόμηση της ε, ειρήνης και της ανάπτυξης είναι πάρα πολύ σημαντικό οι γυναίκες να βρίσκονται σε θέσεις λήψης αποφάσεων ώστε να επιτευχθεί η ειρήνη και να διατηρηθεί στις χώρες. Και η υπηρεσία εξωτερικής δράσης καταβάλει προσπάθεια ώστε να βελτιωθεί η θέση της γυναίκας. Ένα τελευταίο μέσο, όργανο, που θέλω να αναφέρω είναι το Ευρωπαϊκό Όργανο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που ασχολείται ιδιαίτερα με το θέμα της προστασίας των γυναικών και των κοριτσιών. Επιθυμούμε Επίσης να υπογραμμίσουμε το βασικό θεμελιώδη ρόλο των πολιτικών κομμάτων για να υπάρξει μια πραγματική αλλαγή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα το ρόλο έχει η συγκήτρια. Ευχαριστώ πολύ για τα επικοδομητικά σχόλια και προσβλέπω στη συνέχεια να περιλάβω όλα τα σχόλια ώστε να έχουμε μια έκθεση που θα γίνει δεκτή ομόφωνα. Θα ήθελα δύο, σχόλια, δύο σημεία να σχολιάσω. Στην παράγραφο 3, εκεί που λέω όπου είναι ε, ορθό ή κατάλληλο. Αναφέρομαι στα ε, συστήματα, τα εκλογικά, διότι σε κάποια εκλογικά συστήματα έχουν προβλεφθεί ποσοστώσεις, ε, σε άλλα όχι. Ίσως μπορούμε να βρούμε μια καλύτερη διατύπωση για να μην δίδουμε την εντύπωση ότι αφορά όλα τα κόμματα και όλους τους φορείς. Στο άλλο σημείο, για τρεις συνεχείς θητείες να υπάρχει ισόποση συμμετοχή ανδρών και γυναικών. Αυτό για τους εξή λόγους. 50% θα πρέπει να είναι άνδρες και 50% γυναίκες. Αλλά στην Επιτροπή Γυναικών, παραδείγματο χάρη, θα πρέπει να έχουμε τον ίδιο αριθμό ανδρών και γυναικών. Εδώ έχουμε Ε, άνδρα πρόεδρο και δεν θέλουμε να τον αλλάζουμε κάθε χρόνο και να αντικαθίσταται από μια γυναίκα. Άρα λοιπόν, γι' αυτό αναφέρω τρεις διαδοχικές θητείες, ώστε να γίνεται μια εναλλαγή ανδρών και γυναικών τόσο στο Προεδρείο όσο και στη σύνθεση. Ε, για να υπάρξει αυτή η ισότητα και να καταπολεμηθεί η διάκριση σε όλες τις επιτροπές. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και ερχόμαστε και κλείνει το σημείο μάλλον αυτό και πάλι οι προθεσμίες. Σήμερα έχουμε 20 Δεκεμβρίου. Στις 3 το απόγευμα είναι η τελευταία προθεσμία για υποβολή τροπολογιών. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στη συνεδρίαση της 25ης-26ης Ιανουαρίου και θα έρθει στην Ολομέλεια του Μαρτίου η έκθεση. Τελειώσαμε λοιπόν με το σημείο 14 και περνούμε στο σημείο 18 που είναι το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Μεταφορά στο Εθνικό Δίκαιο και εφαρμογή της Οδηγίας του Συμβουλίου 2004, 113 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών. Η κυρία Ζήτα Γκουρμάη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε, αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα αν κρίνει κανείς από την παρουσία των μελών στην αίθουσα. Βέβαια είναι και δικό μου λάθο, γιατί έπρεπε να το συζητήσουμε τον Νοέμβριο. Αλλά ήμουν στο Τόγκο, πρόεδρος εκεί στη Σύνοδο. Και βέβαια αφού ήμουν στην Αφρική δεν μπορούσα να είμαι εδώ. Και επειδή είμαι υπεύθυνη, υπεύθυνο άτομο στη λήψη αποφάσεων, ε, είπα να είμαι εγώ παρούσα. Όχι επειδή δεν έχω εμπιστοσύνη στους συναδέλφους, αλλά ήθελα να είμαι εγώ παρούσα. Ευχαριστώ πολύ την Άντζελα λοιπόν που με αντικαθέστησε τότε. Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον θέμα και μας δίνει, μάλλον μπορεί να χρησιμεύσει ως πρότυπο, ως μοντέλο. Η Κομισιόν είναι επιφυλακτική και θέλω να μάθω ποιος εκπροσωπεί εδώ την Κομισιόν. Μάλλον κανείς δεν μου δίνει σημασία τώρα. Λοιπόν, διαπίστωσα ότι τούτο είναι ένα θέμα το οποίο επηρεάζει την καθημερινότητά τους άνδρες και γυναίκες. Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις υπηρεσίες διότι έχουμε το έγγραφο στις 23 γλώσσες και υπάρχει λοιπόν ίση μεταχείριση στο θέμα αυτό. Θα είμαι πολύ σύντομη στο σχολιασμό, διότι σίγουρα έχουμε και άλλα θέματα στην ημερησία διάταξη. Ευτυχώς όμως έχουμε λίγο χρόνο και μπορείτε βεβαίως να βρείτε αυτό το έγγραφο εργασίας και online και σίγουρα θα είχατε όλη την ευκαιρία να το διαβάσετε και γι' αυτό προτιμώ να ακούσω τις δικές σας σκέψεις παρά να σας παρουσιάσω εγώ μακρηγορώντας το κείμενό μου. Διότι μιλάει από μόνο του ή τουλάχιστον αυτό ελπίζω. Ε, να τονίσω λοιπόν ένα-δύο σημεία. Καταρχήν, είμαι υπεύθυνη για τη συνολική αξιολόγηση της οδηγίας του Συμβουλίου 2004-113. Ωστόσο, αυτό δεν είναι μια αποστολή ρουτίνας. Δεδομένου ότι υπάρχει η απόφαση τεστ άσο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη συντάξει μια έκθεση για το πώς εφαρμόζεται η οδηγία αυτή στις χώρες μέλη. Και η έκθεσή μου και το ψήφισμα θα βασίζεται στο έγγραφο αυτό. Δυστυχώς η έκθεση αυτή δεν είναι ακόμα έτοιμη. Καθυστέρησε, αναβλήθηκε πολλές φορές και προβλέπεται να είναι έτοιμη στο τέλος του έτους. Αν κάποιος είναι εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα να μάθω να μας πει πότε θα γίνει, ότι είμαστε πια στα τέλη του έτους αυτού. Αυτή η καθυστέρηση ήταν κατανοητή καταρχήν, δεδομένου ότι υπήρχε η τεστά case, η περίπτωση αυτή. Αλλά τώρα προτρέπω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα πια και την παρακαλώ να παρουσιάσει την αξιολόγησή της το ταχύτερο δυνατό. Και αυτό είναι σημαντικό διότι έχουμε μια Ευρώπη η οποία που είναι εντελώς διαφορετική. Οι άνθρωποι αισθάνονται ότι δεν τους φροντίζουμε. Δεν μεριμνούμε για αυτούς. Ενώ από την άλλη κάποιοι είναι έτοιμοι να κινητοποιηθούν και να κάνουν κάτι, δεν ξέρουν πώς να δράσουν. Και ε, αυτά ξεκίνησαν το, το Δεκέμβριο του 2010. Έτσι, πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να έχω και το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ τώρα υπάρχουν πολύ σημαντικά σημεία της οδηγής που απαιτούν την προσοχή μας αμέσως για να προκληθεί μια συζήτηση στην Επιτροπή μας και να δω πώς, ποια είναι η αντιμετώπιση σας ως προς την οδηγία και τις επιπτώσεις της περίπτωσης τεστ ασά. Τούτο σημαίνει ότι έπρεπε να βασίσω το έργο μου όχι στην έκθεση της Κομισιόν, αλλά στην έκθεση για τις διακρίσεις των φύλων ε, την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Νομικών Εμπειρογνωμών του Ιουλίου του 2009. Λοιπόν, αυτό το έγγραφο εργασίας είχε την πρόθεση να δώσει μια γενική περιγραφή ως προς την εφαρμογή της οδηγίας και να υπογραμμίσω τις απόψεις μου, να προβάλλω τις απόψεις μου για τα προβλήματα και τις πιθανές λύσεις στο μέλλον. Και γιατί. Γιατί ήθελα να αποδείξω προς την Επιτροπή ότι βρισκόμαστε εδώ για να συνεργαστούμε. Αυτή η έκθεση επηρεάζει και άλλες οδηγίες. Βλέπω καταρχήν κάποιες θετικές εξελίξεις. Ε, υπάρχει μία μεταστροφή για το βάρος απόδειξης. Ότι δηλαδή δεν έχει γίνει παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Αυτή η αρχή έχει εφαρμοστεί στα περισσότερες εθνικές νομοθεσίες. Δυστυχώς δεν καλύπτονται όλα τα κριτήρια σε όλες τις χώρες μέλη. Ένα από τα αποτελέσματα της οδηγίας είναι ότι αυτή τη στιγμή πλειοψηφία των χωρών μελών ε, ρυθμίζουν το θέμα των διακρίσεων σε σχέση με την ε, εγκυμοσύνη και τη μητρότητα. Ε, διότι υπήρχαν τέτοια προβλήματα που συνδέονταν με θέματα στέγασης ε, κλπ. Και επίσης υπήρχαν ε, σημαντικές δυσκολίες νομικής φύσεως σε θέματα δικαιώματος αναπαραγωγής της γυναίκας κλπ. Η ενσωμάτωση ε, της κοινοτικής νομοθεσίας στην εθνική δεν έχει ολοκληρωθεί, σε πολλές περιπτώσεις έχει καθυστερήσει. Πολλές φορές υπάρχουν μινιμαλιστικές προσεγγίσεις και σοβαρές παρεκκλήσεις όταν ερχόμαστε στην εφαρμογή και την υλοποίηση ε, της οδηγίας. Ένα άλλο θέμα όπου υπάρχουν ακόμα σοβαρέ ελλείψεις είναι ο θυλασμός, τα δικαιώματα που προκύπτουν από αυτό. Είναι ενδιαφέρον να υπογραφμίσουμε το θέμα και της ε, ε, σεξουαλικής απειλής ε, τόσο στο χώρο του σχολείου όσο και στο χώρο της εργασίας της εχροσανικής παρενόχλησης και την εξάλληψη των στερεοτύπων. Ε, είναι πολύ σημαντικό να ε, ξεκαθαρίσουν οι διαδικασίες ε, για τις παραβιάσεις και η θέσπιση βάσης δεδομένων για περιπτώσεις τέτοιων παραβιάσεων, ώστε να προστατευτούν τα θύματα τέτοιων διακρίσεων. Όταν ερχόμαστε στα εθνικά όργανα προστασίας της ισότητας, χρειάζεται μια καλύτερη εικόνα για το πώς αυτοί εκπληρώνουν την αποστολή τους. Και το τέταρτο σημείο που αναφέρω συνθέεται στην Test Asha Case. Το άρθρο 5.1, όπως όλοι γνωρίζουμε τις οδηγίες, ε, προσφέρει τη δυνατότητα ε, μάλλον ε, προβλέπει να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση της ισότητας των δύο φύλων στην καταβολή αποζημιώσεων κλπ. Με βάση λοιπόν το άρθρο 5.1 οι χώρες μέλη θα έπρεπε μέχρι το Δεκέμβριο του 2007 να Ε, να εφαρμόσουν ακριβώς αυτή τη διάταξη στις περιπτώσεις εκείνες καταβολής αποζημιώσεων όπου η διαφορά του φύλου έφερνε σε υποδέστερη θέση το θύμα. Ε, υπήρχε βεβαίως η δυνατότητα παρέκκλησης και όλες οι χώρες μέλη έκαναν χρήση αυτής της δυνατότητας παρέκκλησης. Την 1η Μαρτίου του 2011 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, έθεσε εκτός ισχύως αυτή την δυνατότητα απόκλησης, παρέκκλησης από μετά την 31 του 2011. Τούτο σημαίνει ότι το θέμα των αποζημιώσεων καθίσταται ακόμα πιο πολύπλοκο. Ως βουλευτής αυτό που με ενδιαφέρει είναι το συμφέρον των πολιτών, που στην περίπτωση μας είναι καταναλωτές. Αν σκεφτούμε την αγορά, οι μελέτες σαφώς δείχνουν ότι άμεση αύξηση των αποζημιώσεων από ασφάλεια ζωής πρέπει να αναμένεται ιδιαίτερα για τις γυναίκες, υπέρ των γυναικών. Υπάρχει λοιπόν, πρέπει λοιπόν να αναζητηθεί μια πολύ λεπτή ισορροπία. Προτιμώ η ίδια η αγορά να αναπτύξει μια πιο σύνθετη μέθοδο παρά να αυξηθούν οι τιμές. Αλλά δεν φαίνεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ο κλάδος λοιπόν των ασφαλιστικών ε, δεν θα πρέπει να αναλάβει αυτό το ρόλο, δεν είναι αυτός ο στόχος μου. Πρέπει λοιπόν ένα βασικό ερώτημα να απαντηθεί. Άνδρες και γυναίκες βρίσκονται στην ίδια θέση ως προς την ασφάλεια ζωής ή είμαστε διαφορετικοί. Τα στοιχεία δείχνουν ότι σε πολλές περιπτώσεις, ας πούμε το προσδόκιμο, στο προσδόκιμο ζωής, είμαστε σε διαφορετική θέση. Διαφορετική λοιπόν, διαφοροποιημένη μεταχείριση στην ασφάλεια ζωής ε, μέχρι στιγμής ε, τουλάχιστον και μιλάω για τα τελευταία 100 χρόνια ε, θεωρείται ότι δεν υπήρχαν διαφοροποιημένες ε, θέσεις. Μπορεί όμως ο κλάδος να χρησιμοποιήσει αυτή τη διάσταση της διαφοράς των δύο φύλων ώστε να καθορίσει διαφορετικά κριτήρια. Επίσης είναι πολύ σημαντικές οι κοινωνικές συνέπειες από, την ενδεχό, από το ενδεχόμενη αύξηση του κόστους καθώς αυξάνονται, αυξάνεται και η ζήτηση από πλευράς καταναλωτών. Είναι βέβαιο όλα αυτά θα έχουν τις επιπτώσεις τους τόσο στις ιδιωτικές συντάξεις όσο και στις αποζημιώσεις. Και αυτό λαμβάνοντας υπόψη την όλη συζήτηση που γίνεται σήμερα στην Ευρώπη σε σχέση με το ύψος των συντάξεων κλπ. Η απόφαση είχε αναδρομική ισχύ και αρχίζει από την 31η ε, Δεκεμβρίου 2007. Υπήρχε βεβαίως μια σύντομη μεταβατική περίοδος και για να αποφευθούν μελλοντικές διαφωνίες και συγκρούσεις έπρεπε να διασφαλιστεί η νομιμότητα ως προς την εφαρμογή και αυτό είναι πρώτης προτεραιότητας και για τους καταναλωτές. Να είμαστε ειλικρινείς αγαπητοί συνάδελφοι. Αν ο μπει σε δύσκολη θέση ο κλάδος των ασφαλιστικών εταιριών, ποιος θα πληρώσει σε τελευταία ανάλυση εμάς τους καταναλωτές. Η Κομισιόν δηλώνει ότι κατά την άποψή της δεν χρειάζεται μια τροποποίηση της νομοθεσίας. Επίσης η Επιτρόπος Ρέντινγκ είπε ότι η εφαρμογή κατευθυντηρίων γραμμών ή υπό τη μορφή μιας σύστασης θα εκδοθεί το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα. Ακόμα περιμένουμε. Για μένα όμως είναι σαφές ότι χρειάζεται νομική βεβαιότητα χωρίς αμφισημίες και αυτό είναι κατεπήγον. Είναι ε, αμφισβητήσιμο αν αυτές οι μη δεσμευτικέ κατευθυντήριες γραμμές που πρόκειται να εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι απολύτως ικανοποιητικές. Θα πρέπει να δοθεί λοιπόν περαιτέρω προσοχή στην ανάγκη της προσαρμογής της υπάρχουσας νομοθεσίας. Βεβαίως δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά αν δεν θέλει η Κομισιόν να δράσει. Αλλά είναι πολύ η κίνδυνη. Διαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία η οδηγία για την οποία συζητούμε θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβει υπόψη το, την όλη αυτή νομοθεσία. Πιστεύω ότι το έργο μου δεν είναι one woman show. Παρουσιάζω λοιπόν το σχέδιο έκθεσης και θα ήθελα να μάθω τις απόψεις όλων. Και επειδή μοιράστηκα μαζί σας ακριβώς τις δικές μου απόψεις σε σχέση με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Θα ήθελα τώρα να ακούσω και τις δικές σας ε, απόψεις και τα σχόλια και ευτυχώς έχω εδώ την Αντιπρόεδρο Ματέρα. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ. Είχαμε ήδη μια πολύ καλή συζήτηση μαζί σας και το ίδιο ισχύει και για την όλη αξιολόγηση της οδηγίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας εύχομαι όλους καλά Χριστούγεννα. Δεν είναι mission impossible, δεν είναι μια αδύνατη αποστολή αυτή που πρόκειται να αναλάβουμε. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Όπως είπατε, δεν έχουμε και πολλά μέλη παρόντα. Έχω όμως μια ερώτηση για όσα είπατε και όσα έχετε γράψει βέβαια. Στο τέλος της εκθέσης σας έχετε ένα κατάλογο συμπερασμάτων, συστάσεων μάλλον. Λέτε τι πρέπει να γίνει. Έχετε όμως έχετε κάποια πιο συγκεκριμένη ιδέα. Αναμένουμε βέβαια την έκθεση της Κομισιόν. Αλλά μήπως και εσείς έχετε σκεφτεί λίγο περισσότερο τι πρέπει να γίνει συγκεκριμένα όμως. Ο λόγος στην Κομισιόν καταρχήν. Ευχαριστώ. Όπως γνωρίζετε η Κομισιόν ε, έχει προβεί σε διαβουλεύσεις μετά την αποφάση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου με όλους τους ενδιαφερόμενους. Με τους εκπροσώπους των καταναλωτών, τους ασφαλιστές και τα κράτη-μέλη. Η αντιπρόεδρος κυρία Ρέντινγκ ε, αμέσως άλλωστε ε, ανέλαβε τη δέσμευση μέχρι το τέλος του χρόνου να υιοθετήσει κατευθυντές γραμμές για να διευκρινίσουμε τα πιο, τις πιο σημαντικές πτυχές που θίγει η απόφαση του Δικαστήριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να επιτραπεί σε όλους έγκαιρα να την θέσουν σε εφαρμογή αυτή την απόφαση. Αυτές οι κατευθυντές γραμμές πράγματα θα υιοθετηθούν πριν το τέλος του χρόνου, μάλλον αύριο. Οπότε ε, η δέσμευση να υιοθετηθούν ε, μέσα στον ένα χρόνο που έδωσε ως προθεσμία το δικαστήριο ε, θα γίνει σεβαστή. Ευχαριστώ. Okay. Πολύ καλά, λέει ο Πρόεδρος. Και πάλι έχετε το λόγο, έχει το λόγο η ε, δύο γυναίκες έχουμε εδώ και τον Πρόεδρο, ευτυχώς. Έχω μια ερώτηση. Αυτό το έγγραφο θα είναι έτοιμο αύριο και είναι η τελευταία μέρα συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και εμείς χρειαζόμαστε κάποιες διακοπές. Οπότε ας μας σεβαστεί λίγο η Κομισιόν. Γιατί δεν ήταν δυνατόν ε, να μας υποβάλουν τις κατευθείαν γραμμέ λίγο πιο νωρίς. Αυτό το έγγραφο εδώ ήταν έτοιμο μέσα Νοεμβρίου. Δηλαδή εγώ σεβάστηκα πλήρως την Κομισιόν να της δώσω τη γνώμη μας και ε, ε, χαίρομαι που βοήθησαν και οι συνάδελφοι. Η Κομισιόν τελικά δεν ενδιαφέρεται για το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, λυπάμαι που το λέω, αλλά ε, εμάς η γνωμοδότησή ήμασταν έτοιμοι από μετά μέσα Νοεμβρίου και κανένας δεν μου ζήτησε και τη γνώμη μου προσωπικά. Δεν ξέρω αν είχατε επαφή με την Άστρεντ ή με τις υπόλοιπες, αλλά εγώ δεν πήρα ούτε ένα έγγραφο, δεν πήρα καν πρόσκληση όταν το συζητήσατε ως ενδυνάμει εισηγήτρια. Τι είδους συνεργασία θέλετε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να το αντιληφθείτε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πλέον ισχυρότερο από ποτέ. Θα πρέπει να μας σέβεστε ως εκπροσώπους των Ευρωπαίων πολιτών. Και ετοιμάσαμε αυτό το έγγραφο με την ομάδα μας έγκαιρα για να δείξουμε ότι είμαστε και υπεύθυνοι. Και τώρα μου λέτε σε τρεις φράσεις ότι διαβουλευθήκατε. Ε, και λοιπόν Πού είναι το feedback των μελών. Εγώ ξέρω ποιο ήταν το feedback των ασφαλιστών. Ε, γιατί έχουν κάνει μελέτες. Το λάβατε υπόψη σας. Όχι. Δεν το λάβατε. Γιατί η μελέτη δεν είναι έτοιμη. Η Κομισιόν πρέπει να μας σέβεται. Να σέβεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και κύριε Πρόεδρε, μια και κάνατε ένα ερώτημα, θέσατε ένα ερώτημα. Εγώ ε, σας παρέθεσα τις σκέψεις μου και ελπίζω ότι θα με βοηθήσετε για τα περαιτέρω βήματα. Μπορείτε να γράψετε μια επιστολή ως πρόεδρος και να λέτε ότι 20 Δεκεμβρίου και δεν έχουμε πάρει ακόμα τίποτα. Πώς μπορούμε να συνεργαστούμε την Κομισιόν αν τα πράγματα διεξάγονται με αυτόν τον τρόπο. Και και ε, περιμένουμε και άλλα κείμενα από την Κομισιόν στο μέλλον. Τι θα γίνει, με τον ίδιο τρόπο θα τα χειριστούμε. Mm. Υπάρχει μια ηθική κρίση στην Ευρώπη και θα πρέπει να δείξουμε στους πολίτες ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι και κάνουμε κάτι εξ ονόματός τους. Χαίρομαι που το έγγραφο θα είναι έτοιμο αύριο, αλλά <laughs> όμορφο αυτό το ότι στηρούμε την πλασμία των οσέτους, αλλά δυστυχώς πριν την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου δεν πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να αντιδράσουμε δεδομένου ότι όλοι μας χρειαζόμαστε ε, διακοπές τα Χριστούγεννα. Ελπίζω ότι στο μέλλον η Κομισιόν θα κάνει τα πράγματα καλύτερα. Δεν είμαστε μαριονέτες. Είμαστε σοβαροί στη λήψη αποφάσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ωραία. Κανεί άλλο δεν θέλει το λόγο νομίζω αυτή τη στιγμή. Ωραία. Να θεωρήσω ότι η λίγη συζήτηση για αυτό το ζήτημα. Να σας πω δύο λόγια για το χρονοδιάγραμμα. 26 Φεβρουαρίου, 28 Φεβρουαρίου, συγγνώμη, ε, θα συζητηθεί η έκθεση αυτή. 1η Μαρτίου η προθεσμία για τροπολογίες, 12 το μεσημέρι. Η... Θα ψηφίσουμε στις 27 Μαρτίου, εμείς εδώ, και δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχουμε αποφασίσει πότε θα συζητηθεί από την Ολομέλεια. Περνάμε στο σημείο 16. Σημεία 16 και 17 συγκεκριμένα, νομίζω μπορούμε να τα συζητήσουμε μαζί, γιατί σχετίζονται και βέβαια είναι και η ίδια η συγγήτρια. Αν κανείς δεν έχει αντίρρηση λοιπόν, να τα δούμε μαζί τα σημεία 16 και 17. Κύριε Ματέρα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως και η συνάδελφος ε, Τζίτα, ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα θέματα ε, γι' αυτό ακριβώς μαζικά συμμετέχουν και παρίστανται οι συνάδελφοι. Εν πάση περιπτώσει έχουμε τον πρόεδρο, έχουμε εξαιρετική, είμαστε εξαιρετική συντροφιά. Ε, ε, ε, λοιπόν, ε, εξ ονόματο τη Επιτροπή ε, Γυναικών είμαι υπεύθυνη για τη, υπεύθυνη για τη σύνταξη γνωμοδότηση. Γνωρίζετε ότι η διάσταση φύλου είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και η Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, εξετάζει κατά πόσον γίνεται σεβαστή η διάσταση αυτή ε, στον προϋπολογισμό και στις γραμμές του προϋπολογισμού. Ε, η πρώτη μου ε, απαλλαγή αφορά τον γενικό προϋπολογισμό ενώ στη δεύτερη γνωμοδότησή μου ε, κυρίως ασχολούμαι με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φίλων στο Βίλνιους. Όσον αφορά τον γενικό προϋπολογισμό δεν έχω πολλά πράγματα να πω και θα δείτε άλλωστε ότι και η γνωμοδότηση είναι δύο-τρεις παράγραφοι όλοι και όλοι. Ε, απλώς ε, την ε, ανάγκη ε, ο έλεγχος του προϋπολογισμού που εμπεριέχει τη διάσταση του φύλου να αποτελεί προϋπόθεση για την προπαρασκευή ενός προϋπολογισμού που εμπεριέχει και αυτό στη διάσταση του φύλου. Ε, στην άλλη γνωμοδότηση που είναι και μακρύτερη αφορά τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φίλων στο Βίλνιους στον, ε, ε, στο ε, κεφάλαιο 2, στον τίτλο 2 μάλλον, δαπάνες υποδομών και λειτουργίας, δεσμεύτηκε ένα ποσό ύψους 195.000 ευρώ. Και αυτό γιατί μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου του 2011 ε, ε, υπήρχαν έξοδα ενοικίασης, μάλλον δεν υπήρχαν έξοδα ενοικίασης γιατί η, η λιθουανική κυβέρνηση ε, ήταν αυτή η οποία κάλυψε τα έξοδα ενοικίασης. Όσον αφορά τώρα τον τίτλο 3, λειτουργικές δαπάνες, παρατηρούμε ότι υπάρχει ένα ποσό ύψους 220.000 ευρώ ε, το οποίο δεσμεύτηκε λόγω ανεπαρκού απορρόφηση για λειτουργικά έξοδα λόγω ε, της δυσκολίας που είχε το Ινστιτούτο αυτό να προσλάβει προσωπικό με προσόντα ε, ικανά να αντιμετωπίσουν τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου αυτού. Υπήρχαν λοιπόν και νέες θέσεις ε, όσον αφορά τους εμπειρογνώμονες ε, που θα ε, κάνουν έρευνα λοιπά Και που θα διασφαλίσουν την σωστή λειτουργία του Ινστιτούτου στο μέλλον. Σε σχέση πάντα με την γνωμοδέτησή μου, υπογραμμίζω ότι το Ινστιτούτο θα πρέπει να σημειώσει ποια είναι ε, τα προσκόμματα τα οποία έχει αντιμετωπίσει στη διάρκεια της λειτουργίας του έτσι ώστε με σαφήνεια αλλά και διαφάνεια να λειτουργήσουμε και εμείς και εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ας πούμε να έχουμε την απαραίτητη πληροφόρηση. Ε, εδώ θα ήθελα και εγώ να ε, αναφερθώ στο χρονοδιάγραμμα γιατί η 9η Νοεμβρίου, ε, συγγνώμη, Ιανουαρίου του 2012, δηλαδή αμέσως μετά την επανέναρξη των ε, εργασιών μετά τις ε, διακοπές είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Πρόκειται για δύο γνωμοδοτήσεις ε, οι οποίες ήταν μεν απλές αλλά και πολύ σημαντικές κατά την άποψή μου. Δηλαδή αφορούσαν θέματα σημαντικά. Ε, και ε, ε, πρέπει οπωσδήποτε να λειτουργήσει σωστά αυτό το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φίλων στο Βίλνιους. Αυτά. Νομίζω ότι με τις, εργα... με τις δικές μου εκθέσεις ολοκληρώσαμε και τις εργασίες μας. Χαίρομαι που έχουμε έναν πρόεδρο που είναι και άνδρας και ικανός και δραστήριος και παρόν και μακάρι να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας πάντα ε, με τον ίδιο τρόπο. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ, που είστε αυτός που είστε και που κάνετε αυτή τη δουλειά που κάνετε τόσο καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, έβγαλε τα ακουστικά μου μισό λεπτό, αλλά άκουσα τι λέγατε. Ένα δευτερόλεπτο. Σας άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και εξάλλου μαθαίνω και Ιταλικά, μην ξεχνάτε. Exactly, our Hungarian translator said that probably... Ναι, ενδεχομένω ε, καταλαβαίνετε καλά Ιταλικά, αυτό μου είπανε και εμένα. Okay. So. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ακόμα και ένα θέμα το οποίο είναι τόσο, τόσο σημαντικό και ενδιαφέρον ε, και έτσι ψηρέουν τα πλήθη για να το ακούσουν, δηλαδή για τον γενικό προϋπολογισμό ε, αξίζει να μας απασχολήσει. Είναι γεγονός βέβαια ότι και η Μπάρμπαρα σαν νέα ε, νέα και δραστήρια έχει ε, επιβεβαιώσει την παρουσία της ε, σε αυτό τον ανδροκρατούμενο τομέα της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμών. Υπάρχει μία πρόταση επισημαίνει ότι ένας έλεγχος του προπολογισμού που εμπεριέχει τη διάσταση του ε, φύλου αποτελεί προϋπόθεση για την προπαρασκευή ενός προϋπολογισμού που εμπεριέχει τη διάσταση του φύλου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ε, ε, πραγματικά αντικατοπτρίζει την άποψη που έχουμε εμείς για την συνεργασία. Όσον αφορά τώρα το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, είναι ένα Ινστιτούτο το οποίο εκπονεί πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες μελέτες ε, ή τέλος πάντων έχει το δυναμικό για να εκπονεί τέτοιε μελέτες ακόμα δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο ε, υπάρχουν κάποια προβλήματα όσον αφορά το προϋπολογισμό ε, του Ινστιτούτου είναι σαφές ότι πρέπει να δουλέψει σωστά Χθες μόλις διάβασα μια έκθεση σχετικά ε, με την διάσταση του φύλου στην οικονομική κρίση και ε, αυτό με ενδυνάμωσε ακόμα περισσότερο τη θέση μου ε, όσον αφορά την ανάγκη στατιστικών στοιχείων, την ανάγκη δεδομένων ε, για όλα τα θέματα αυτά. Ε, πιστεύω ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ευχαριστούμε τη Μάρβαρα γιατί έκανε πολύ καλή δουλειά, όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση, αλλά κάθε φορά που είναι υπεύθυνη για κάτι, πραγματικά το κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν ε, όλους ε, όσους έκαναν, ε, μας βοήθησαν στη δουλειά μας και τους διερμηνείς. Ευχαριστούμε και εμείς. Και Μιχαήλ, να πω ότι είναι σημαντικό να έχουμε μια ισχυρή παρουσία και είναι πολύ σημαντικό που είσαι εδώ, που είσαι πρόεδρος και που είσαι τόσο ευαίσθητος όσον αφορά τα θέματα που από τη διάσταση του φίλου. Ευχαριστώ. Να υπογραμμίσω μονάχα το γεγονός ότι όπως είπε και η κυρία Ματέρα είναι κρίμα που δεν υπάρχουν πολλές τέτοιες προτάσεις και κρίμα που δεν είχαν μπει κάποια στοιχεία από την αρχή και έπρεπε να μπουν εν είδη τροπολογιών. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ενώσω τη φωνή μου στις ευχές που διατυπώθηκαν προς όλους. Και θέλω να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερος το έργο και την αφοσίωση της Μπάρμπαρα. Έργο, αφοσίωση που επέδειξε στην περίπτωση αυτή και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο κάναμε και πέρσι όταν συζητούσαμε τον προϋπολογισμό ή την απαλλαγή. Θα ήταν καλό να έχουμε εδώ τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων. Γιατί χρειάζονται στοιχεία και μερικές φορές χάνουμε την ε, επαφή με αυτό το Ινστιτούτο. Και είμαι βέβαιη ότι θα έχουν προβλήματα μεταφέροντας το Ινστιτούτο σε κάποιο άλλο κτίριο και ο συντονισμός μεταξύ αυτού και αυτής της Επιτροπής ελπίζω ότι στο μέλλον θα είναι καλύτερος. Ε, το λέω αυτό επειδή ξέρω ότι έχουμε στραμμένο το ενδιαφέρον στην προετοιμασία του νέου Προεδρίου αλλά γνωρίζω αλλά ελπίζω ότι θα έχουμε το χρόνο να καλέσουμε την κυρία Λάμπα και κάποιον άλλον ώστε να διατηρηθεί αυτή η σχέση και ο σύνδεσμος με την Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή, ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε το τι συμβαίνει. Γιατί έχουμε συμφωνήσει ότι τουλάχιστον μια φορά το χρόνο θα έχουμε μια τέτοια συζήτηση. Και έχω την εντύπωση ότι Ειδικά όταν συζητούμε προϋπολογισμό ή απαλλαγή, καλό είναι να συζητάμε μαζί τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Συμφωνώ μαζί σας. Θα λάβω υπόψη αυτό την πρόταση, είναι καλή πρόταση και θα το περιλάβουμε στο σχεδιασμό μας. Υπάρχει κανείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δυστυχώς δεν έχω όνομα, αλλά θα θέλαμε να ακούσουμε και τις σοφές απόψεις της Κομισιόν. Όχι. Όχι, δεν έχουμε. Δεν θέλει κανείς να πει τίποτα. Όχι, δεν θέλει. εντάξει. Στην περίπτωση αυτή δίνω το λόγο στην Σύγετρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, συμφωνώ πολύ με την πρόταση τη ε, συναδέλφου Μπάουερ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε, να καλέσουμε εδώ ε, κάποιον υπεύθυνο του Ινστιτούτου αυτού ε, έτσι ώστε να ε, συζητήσουμε σε βάθος κάποια θέματα. Δυστυχώς και σήμερα δεν έχουμε πολλούς συναδέλφους ε, για να κάνουμε έτσι μια συζήτηση σε βάθος. Τα θέματα του προϋπολογισμού θεωρούνται λίγο δύσκολα. Εγώ όμως θα ήθελα να πω ότι ε, τα θέματα του προϋπολογισμού ε, τα θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά ε, και μάλιστα όπως μου έλεγε και ο επικεφαλής αντιπροσωπείας μου ο Μάριο Μάουρο μη φοβάσαι προχώρα και ε, μελετώντας και προσέχοντας ε, θα πας ε, πολύ μακριά και θα τα καταλάβεις όλα. Εγώ λοιπόν σιγά σιγά απέκτησα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα θέματα αυτά και πραγματικά θα ήθελα να στηρίξω, να μεταδώσω μάλλον το ενδιαφέρον αυτό και στους συναδέλφους και να στηρίξω την πρόταση της συναδέλφου Μπάουερ. Eh, eh, Ευχαριστώ πολύ. Άρα ολοκληρώσαμε και τη συζήτηση αυτή. Να ξαναδούμε την, το χρονοδιάγραμμα και για την ε, έκθεση, για την γνωμοδότηση αυτή. Τροπολογίες, υποβολή τροπολογιών σήμερα μέχρι τις 3 το απόγευμα. Θα ψηφίσουμε στις 16 Ιανουαρίου και η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού θα μελετήσει το θέμα αυτό στις 28 Μαρτίου. Σήμερα πάντως λίγη η προθεσμία για τις τροπολογίες. 19 λοιπόν, σημείο 19 της ημερησίας διατάξεως, υπό τα διάφορα υπάρχει κάτι. Όχι, επομένως προχωρούμε. Σημείο 20, προσεχή συνεδρίαση, θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες 25 και 26 Ιανουαρίου 2012. Ε, Με την ευκαιρία αυτή λοιπόν Ε, και μια και κοντεύουν τα Χριστούγεννα και θα ξεκουραστούμε όλοι, να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, ευτυχές στο νέο έτος και οι ευχές ισχύουν και για τους διερμηνείς βεβαίως και οι διερμηνείς ευχαριστούν τον Πρόεδρο. όλους όσους συμμετέχουν και βοηθούν στις εργασίες της Επιτροπής. Ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα να ξεκουραστούν. Αξίζετε την ξεκούραση αυτή, την κερδίσατε έτσι με τον υδρότα του προσώπου σας και να ξανάρθετε τον Ιανουάριο πιο δυνατή έτσι ώστε να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε όλα τα ζητήματα τα οποία θα έχουμε ε, στις νέες μας ημερησίες ε, διατάξεις.